Right, if we could uh, calm down, everybody, thank you very much. Uh, I'll run very quickly through the first formalities, first the adoption. Καταρχήν πρέπει να υιοθετήσουμε την ημερησία διάταξη και θεωρούμε ότι έχει γίνει αποδεκτή. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι στις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς και ε, θα πάμε μέχρι τις 6 και 4 διότι πριν από την ακρόαση για την ε, ε, οικονομική διακυβέρνηση που θα ξεκινήσει στις 3 ο Επίτροπος Μπανιέ θα μας παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες που θα έχουν υιοθετηθεί εκείνο το πρωί σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες. Γι' αυτό και δέχτηκα να έρθει κατευθείαν από τη συνεδρίαση και να είναι ο πρώτος, η πρώτη στους οποίους θα απευθυνθεί με, μόλις τελειώσει τη συνέντευξη τύπου. Σήμερα μετά από την ανταλλαγή από, ε, απόψεων με τον κύριο Ρέιντερς θα ε, συζητήσουμε την έκβαση του τριμερούς διαλόγου, πράγμα το οποίο πρέπει να υιοθετηθεί από την Επιτροπή ε, σύμφωνα με, την, ε, τον νέο κανονισμό και μετά ε, τους κανόνες σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ που προβλέπεται στο σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως. Με αυτά χαιρετίζω τον Didier Reinders πρόεδρο του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ, ο οποίος είναι έλγος ε, ε, αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και πρώην ευρωβουλευτές. Ε, θέλω να τον χαιρετήσω ιδιαίτερα θερμά, διότι από κοινού έχουμε συμμετάσχει σε πολλούς τριμερείς διαλόγους και από τις δύο πλευρές του τραπεζιού από όταν ξεκίνησε η Βελγική Προεδρία και ευχαριστώ τον Διδιέ ο οποίος προώθησε τον ε, τριμερή διάλογο για να μπορέσουμε να έχουμε ε, ε, καλή έκβαση. Ο κύριος Ρέντερ, ευχαριστώ. Ο, όντως με συγχωρείτε που καθυστέρησε. Έχουμε και στο Βέλγιο ορισμένες συζητήσεις, αλλά προσπάθησα από την 1η Ιουλίου να ξεκινήσω και να μπορέσουμε παρόλα τα εσωτερικά μας προβλήματα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον εισηγητή για την ε, χρηματοοικονομική εποπτεία που ήταν δύσκολο θέμα. Κάναμε πολλές συνεδριάσεις από την 1η Ιουλίου και ήταν η πρώτη βασική συζήτηση που ελήφθη στο Στρασβούργο να καθυστερήσουμε την συζήτηση ε, σχετικά με το θέμα αυτό και χαίρομαι που μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και όλους τους παρόντες στην αίθουσα διότι μπορέσαμε όλα αυτά να τα επιτύχουμε ε, σε ένα πνεύμα αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επετεύχθη αυτή η συμφωνία και ελπίζω το Κοινοβούλιο θα επιβεβαιώσει τη θέση του τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Ο κύριος Γκοζές είναι στις πρώτες, ε, ε, στα πρώτα έδρανα σχετικά με ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ίσως δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα όσο με την εποπτεία, αλλά είναι σοβαρό θέμα και θα προσπαθήσουμε μεσοπρόθεσμα να βρούμε μία λύση, διότι πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε όχι μόνο να καταρτήσουμε τους νέους θεσμούς εποπτείας την 1η Ιανουαρίου του επομένου ότι θα υπάρχει μια νέα επιτροπή υπεύθυνη για τους συστηματικούς ε, κινδύνους και να μπορέσει ο Μισελ Μπανιέ να παρουσιάσει τα νέα κείμενα ε, κανονισμών. Ακούσαμε ε, το προσχέδιο αυτή την εβδομάδα ε, σχετικά με το επενδυτικό ταμείο. Καταρχήν όμως η πρώτη προτεραιότητα της Βελγικής Προεδρίας ίσως όχι μόνο στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ αλλά στα πλαίσια της Προεδρίας γενικώ είναι να προωθήσει τα μαθήματα που αποκομίσαμε από την κρίση τα τελευταία δύο χρόνια και ίσως και περισσότερο αναλόγως του αν πάει κανείς από το φθινόπωρο ή από τα πρώτα κρούσματα στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική ελέγχου νομίζω ότι το έχουμε επιτύχει με ορισμένες ρήτρε αναθεωρητικές που αποτελούν πλαίσιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και ελπίζουμε ότι τα νέα θεσμικά όργανα θα αποδείξουν ότι είναι αποτελεσματικά και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και περαιτέρω και να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν ότι σε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια όταν θα κοιτάξουμε τις ρήτρε αναθεώρησης θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορούν να αποφασίζουν πέραν των εθνικών κρατών που γνωρίζουμε σήμερα. Τόσο το καλύτερο αν αυτό αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια των ατόμων που από κοινού έχουμε επιλέξει, αλλά αν χρειαστούν άλλοι, το βασικό είναι να αποκομίσουμε τα σωστά μαθήματα από το μηχανισμό που θα καταρτήσουμε. Γι' αυτό και η Προεδρία του Βελγίου είναι πολύ ευτυχής να διαπιστώνει ότι η πρώτη μας προτεραιότητα ήδη στα μέσα του Σεπτεμβρίου υλοποιείται. Άρα προχωράμε στην ε, ε, ε, χρηματοοικονομική εποπτεία, σωστά και ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες στις ε, συνεδριάσεις που θα λάβουν χώρα στις Βρυξέλλες από αρχές Οκτωβρίου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πρωτοβουλία σχετικά με τα επενδυτικά ταμεία. Θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες αλλά αυτή είναι η πρώτη μου προτελεότητα Δεν έχω να πω άλλα πράγματα σχετικά με την ε, ε, χρηματοοικονομική εποπτεία και τα κείμενα σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω όμως ότι είναι βασικό να συνεχίσουμε συνεχίσουμε με την ίδια αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου και να μπορέσουμε υπό καλές προϋποθέσεις να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα στα πλαίσια αυτά. Θέλω όμως να πω και ε, για άλλα πράγματα, για την φορολογική ολοκλήρωση. Ε, στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου θα υπάρξει στο ΕΚΟΦΗΝ μια νέα συζήτηση αφενός για το πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, να έχουμε δηλαδή καλύτερο φορολογικό συντονισμό και ενοποίηση στην Ευρώπη και να καταρτήσουμε νέους στόχους και ε, νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, να υπάρχει δηλαδή ένα κράτος κοινωνικής αβημερίας που προβλέπεται για το 2020, αλλά ποιες είναι οι διαδικασίες για να το επιτρέψουμε. Στο τελευταίο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ε, λάβαμε αυτές τις αποφάσεις και από 1η Ιανουαρίου θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζονται όμω και άλλα. Ορισμένες κυρώσει. αν χρειαστεί για ορισμένε χώρες οι οποίες έχουν πολιτικές που δεν συνάδουν με την φορολογική ενοποίηση και να κοιτάξουμε αν είναι δυνατόν να έχουμε νέο στόχο για το 2020, αποκινούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο για να υπάρχει μία ισοσκελισμένη φορολογική θέση στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά γιατί με τη νέα αυτή διαδικασία, τη νέα στρατηγική θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να βελτιώσουμε την κοινωνική πρόνοια και να αντιληφθούμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε τις χρηματολογικές αλλαγές. Να στηρίξουμε δηλαδή όλες τις χώρες για να γίνει κάτι τέτοιο και να καταπολεμήσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές. Άρα, στο επόμενο άτυπο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ θα υπάρξει αυτή η συζήτηση. Θα προσπαθήσω να καλέσω και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε να προβούμε σε αυτή τη διοργάνωση. Σας είπα ότι αποφασίσαμε αποφασίσαμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά ε, επιζητούμε και μία νέα διαδικασία. Για συγκεκριμένα θέματα θα επανέλθω. Μετά θα επανέλθω και στην ε, εποπτεία. Στο εκοφήν του τέλους του μηνός πρέπει να προβούμε σε μία ανάλυση να ανταλλάξουμε με απόψεις με τις ε, εταιρείες βαθμολογήσεως και τις rating agencies δηλαδή και να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω με ένα καλό πρόγραμμα στην Ευρώπη όπως αυτό που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Να υπάρχει δηλαδή μία σύγκριση μεταξύ της εξελίξεως στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρώπη. Έχουμε πολλά κοινά ε, για τόσα σημαντικά θέματα που αποφασίζονται στο, Αμερικανικό Κογκρέσο ε, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική εποπτεία και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Μπαρνιέ, τον Επίτροπο, να παρουσιάσει μία σύγκριση όσον αφορά τις εξελίξεις ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και στο Στρασβούργο Θέλω ε, να προσκαλέσω την πρόεδρό σας την κυρία Μπόλς να συμμετάσχει σε μια συζήτηση που θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά κατά τρόπον ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να συζητήσουν αν μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα στην Ευρώπη και ε, να ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Άρα στην άτυπη συνεδρίαση στο τέλος τέλος του μηνός θα καταρτήσουμε και το πρόγραμμα για το G20 και ε, για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα πρέπει να συντονίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων επί του θέματος. Μπορώ να σας πω ναι, και να προεξοφλήσω ότι για τη Βελγική Προεδρία όχι μόνο στα πλαίσια της Προεδρίας της αλλά γενικότερα είναι βασικό να προχωρήσουμε στη ρύθμιση των χρηματαγορών ε, όπως το πράττουμε από κοινού το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσπαθήσουμε να δούμε αν έχουμε έναν ε, καλό ρυθμό πρόοδου σε σχέση με τα άλλα μέρη του κόσμου και ε, την δημοσιονομική οικονομική ολοκλήρωση θυμόμενη ότι το σύμφωνο σταθερότητα και αναπτύξεως δεν προβλέπει μόνο σταθερότητα αλλά και ανάπτυξη άρα η ε, την ε, ε, στρατηγική για το 2020 που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα κοινωνικά θέματα και την κλιματολογική πολιτική. Δεν θα επεκτείνουμε επεκταθώ περαιτέρω στα θέματα αυτά γιατί τα γνωρίζετε. Τα έχουμε συζητήσει από αρχές Ιουλίου επανειλημμένως αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τραπέζι του Συμβουλίου υπάρχουν ορισμένοι φάκελοι οι οποίοι πρέπει να εξελιχθούν, να προχωρήσουν. Και αναφέρουμε στο φορολογικό θέμα, διότι η συζήτηση επί της χρηματοοικονομικής εποπτείας ίσως μας έκανε να ξεχάσουμε ότι έχουμε ορισμένα φορολογικά θέματα σε εκκρεμότητα, όπου πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε την την ε, φοροδιαφυγή και πόσο εις ε, το ΦΠΑ αλλά και γενικότερα να ενισχύσουμε την ε, κοινή δράση για να αποφύγουμε την φοροδιαφυγή διότι σε διάφορους τομείς σκέφτομαι όχι μόνο το ΦΠΑ αλλά και στην αποταμίευση και τη φορολογία της μπορούμε να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την καταπολέμηση κατά της φοροδιαφυγής ή της αποφυγής φορολογίας και θα συζητήσουμε με τον κύριο Σεμέτα, τον αρμόδιο επίτροπο, για να δούμε αν μπορούμε να προωθήσουμε την εναρμόνιση και ολοκλήρωση των πολιτικών μας όσον αφορά τη φορολόγηση της αποταμίευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ορισμένες τρίτες χώρες. Και πιστεύω ότι η κρίση δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτό το βασικό φάκελο της φορολόγησης της αποταμιεύσεως που συζητείται και ακόμη δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά που μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά. Θα ήθελα λοιπόν να, σας, να επίσης και δύο ή μάλλον τρεις απόψει ολοκληρώνοντας και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που θα συζητήσουμε ίσως ήδη στο επόμενο άτυπο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Πρώτον, το πρώτο θέμα αναφέρεται εις ε, την ε, ε, εξέλιξη των λογιστικών προτύπων διεθνώς διότι βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να επηρεάζει τις χρηματαγορές ελέγχοντας τα λογιστικά πρότυπα στους θεσμούς που έχει αρμοδιότητα δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει όντως να παρίστεται στις αποφάσεις συστάσεως ε, ε, και ε, καταρτήσεως ε, ε, των μελών ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και θα πρέπει να μπορέσουμε επίσης να συμμετάσχουμε εις τον οργανισμό που καταρτίζει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Το συζητήσαμε τον κύριο Μπερνιέ, θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά θα ήθελα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσουμε την ίδια απορία. Δεν θέλουμε δηλαδή να διευκολύνουμε τους ε, κανόνες, ε, τους λογιστικούς για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις μας, αλλά για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Να ξέρουμε δηλαδή ε, τι γίνεται εις τους οργανισμούς οι οποίοι καταρτίζουν τα λογιστικά πρότυπα χωρίς να παρεκκλίνουμε από την άποψη που έχουμε σαν Ευρωπαίοι επί του θέματος. Άρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες ομάδες και επίσης έχουμε ανακοινώσει μία συμφωνία των κεντρικών τραπεζών και ε, των ρυθμιστών σχετικά με τη Βασιλεία 3. Δηλαδή τα πρότυπα που αναφέρονται στα ίδια κεφάλαια για, τους για τα τραπεζικά ιδρύματα. Και είχα πει ε, σαν, ε, ε, σαν υπουργός σε εθνικό επίπεδο ότι αντιμετωπίζω αντιφατικά θέματα, δηλαδή ε, πώς θα διευκολύνουμε την, ε, ε, τις πιστώσεις από την τράπεζα, πώς θα αξιολογήσουμε την κατάσταση της τράπεζας. Τα θέματα είναι ίσως αντικρουόμενα και οι βουλευτές μας θέτουν ερωτήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε συνεκτικά να συνδυάσουμε τις, ε, τα ίδια κεφάλαια και τις απαιτήσει τους, τη δυνατότητα πιστοληπτικής ικανότητας ε, και ζήτησα στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ μαζί με τον πρόεδρο της ε, τραπέζης, του Ευρωπαϊκής Τραπέζης του κύριο Τρισέ να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα μαζί. Όχι ένα μετά το άλλο, αλλά να δούμε πώς θα εντάξουμε όλους τους νέους αυτούς κανονισμούς σχετικά με την εποπτεία των ιδίων κεφαλαίων, της πιστοληπτικής ικανότητας και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή όπως σας είπα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και με το Κοινοβούλιο πριν το τέλος του έτους για να ολοκληρώσουμε τις διάφορες οπτικές γωνίες. Τρίτον, Θέλω να πω ότι υπάρχουν και συζητήσεις για την προετοιμασία της επομένης Γενικής Συνελεύσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μιλάμε για τη νέα διακυβέρνηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την ε, νέα καλύτερη εποπτεία σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά πρέπει κάτι να σας πω με ένα παράδειγμα. Προετών ε, αρκετών είχαμε καταρτήσει με τα μέλη του ΕΚΟΦΗΝ ότι θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μόνο μία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την, ε, ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή τουλάχιστον μία έδρα για την Ευρωζώνη και πρέπει να σας πω ότι προσωπικά είμαι πεπισμένος. Το ερώτημα είναι μπορούμε να πείσουμε όλους τους συμμετέχοντες στην Ευρωζώνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή η λύση θα είναι καλή. Διότι αν δεν το πετύχουμε είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε και να βρούμε μια άλλη εναλλακτική λύση. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να το συζητήσουμε στην Ευρώπη και επίσης είναι να καλό είναι να συζητήσουμε διάφορα θέματα και θα δώσω άλλο ένα παράδειγμα, όχι παραπάνω. Είναι φυσιολογικό ότι έχουμε μόνο δικαίωμα βέτο από τις Ηνωμένε Πολιτείε ή στην ε, Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στον οργανισμό ολόκληρο ή όχι. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε σίγουρα περισσότερα, να βελτιώσουμε την καλή διακυβέρνηση του Διεθνούς Αστυνομισματικού Ταμεία και από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και της Ευρωζώνης και να θέσουμε στο τραπέζι διάφορα θέματα, ίσως αντιφατικά, στα οποία διαφωνούμε με τις άλλες πλευρές του κόσμου. Το, θα το συζητήσουμε συζητήσω λοιπόν με ε, τα στελέχη του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και άλλους εταίρους μας για να συζητήσουμε όχι ένα-ένα τα θέματα αλλά όλα τα θέματα μαζί για όλες τις ε, ε, υπήρους. Ξέρω ότι και εσείς και εμείς και η Επιτροπή έχουμε και άλλα θέματα αλλά νομίζω ότι από τη μία πλευρά η εποπτεία και η χρηματοοικονομική ρύθμιση η από την άλλη πλευρά η βελτίωση του ε, κοινωνικού πλαισίου και ε, κάποια συζήτηση σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Διεθνή Οργάνωση για τα Λογιστικά Πρότυπα κτλ. που είναι βασικά. Ε, θέλω να κλείσω και να τελειώσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί κατά τη γνώμη μου αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία στις επόμενες εβδομάδες για την χρηματοοικονομική εποπτεία θα είναι πραγματική επιτυχία. Ε, προσβλέπουμε και σε περισσότερα, αλλά σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας. All right, that's better. Yeah, sorry. I'm confused. I've got too many buttons. Δυστυχώς μπέρδεψα τα κουμπιά. Έχω τόσα πολλά μπροστά μου. Λοιπόν, θα σας αναγνώσω τον κατάλογο των ομιλητών. So, uh, so far, I, I... Philippe Lambert, Peter Skinner, Dirk Epping, Vicky Ford. I coffee. Mrs. Tissan. Mrs. Uh, uh, anybody else? Oh, oh, hang on. Υπάρχει κανείς άλλος, γιατί μπέρδεψα τα χέρια αυτών που θέλουν να μιλήσουν και αυτών που ζητούσαν καφέ. Λοιπόν, να σταματήσουμε και θα αρχίσουμε το Ζαν Πολ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ, καταρχάς ε, θα ήθελα να σας πω ότι οι ανησυχίες τις οποίες αναφέρετε ε, είναι ανησυχίες που έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Να συγχαρώ και εγώ την Προεδρία για την επιτυχία του πακέτου για την εποπτεία ήταν πολύ σημαντική επιτυχία και χαίρομαι πολύ που βλέπω και τη δική σας ενεργό συμμετοχή και στην οδηγία, στον τριμερή διάλογο του Στρασβούργου για το, για το και με τον κύριο Μπαρνιέ και μαζί σας οι τρεις μας καταφέραμε νομίζω να καθορίσουμε το πλαίσιο και να δούμε και τα υποσυζήτηση σημεία. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, α όχι λάθος, μπορεί να γίνεται κάποια στιγμή. Κύριε Πρόεδρε πάντως, ε, προς το παρόν, Ας μην ε, ε, βγούμε από, το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Πάντως και οι συνάδελφοί μου ασχολούνται με πολλά ζητήματα. Πάντως έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και σήμερα το πρωί, νομίζω ότι όπως και την Παρασκευή, λειτουργήσε καλά η Task Force για τις τεχνικές πτυχές. Δύο ζητήματα απομένουν, όπως ξέρετε, το equity και οι τρίτες χώρες. Private equity το πρώτο θέμα, θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουμε στο θέμα αυτό. Και πραγματικά θα είναι πολύ καλό και αποτελεσματικό αν την Τετάρτη στον τριμερή διάλογο καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο για το private equity ώστε να έχουμε πραγματική διαπραγμάτευση για να έχουμε μια συμφωνία, όχι με κάθε τίμημα ή με οποιοδήποτε τίμημα. Αναφέρατε και εσείς τα σχετικά και νομίζω ότι αν προτείνει η Προεδρία και δεν είναι εύκολο βέβαια. Αν η Προεδρία προτείνει ένα κείμενο που περιλαμβάνει τι βασικέ θέσει, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Για τι τρίτε χώρε τώρα ξέρω ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή από τα κράτη-μέλη. Κάθε ένα κάνει τι δικέ του προσπάθειε και εγώ κάνω τι δικέ μου προσπάθειε για να απεμπλακούν τα πράγματα, τουλάχιστον σε μια χώρα την οποία γνωρίζω εγώ καλύτερα από άλλε. Και βέβαια πρέπει κανείς να μιλά, να έχει το θάρρος της γνώμη του και να διαφωνεί ενδεχομένω με τους υπόλοιπου. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι μόνο μιλάνε και είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν πράγματα και πολλές φορές και στις εκλογές ε, βλέπουμε ε, πώς ανταμείβεται ο ημέν και η δέγο. Ε, νομίζω ανήκω και στις δύο κατηγορίες. Και λέω και Πράτο. Θα ήταν δραματικό νομίζω να μην καταλήξουμε σε μια λογική συμφωνία Ξέρουμε ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα και είναι ευαίσθητοι οι συμπολίτε μα. Μπορεί να μην γνωρίζουν τι τεχνικέ λεπτομέρειε. Έχουν δει όμω ε, τι ζημίε είχαμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αν σήμερα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορέσει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε λύσει, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ πώ θα αντιμετωπίσουμε με ηρεμία την Γαλλική Προεδρία του G20 αν θέλουμε να λύσουμε κάποια ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, πρώτα πρέπει να τα καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ γιατί ήταν πολύ αποφασιστικός. Νομίζω ότι προσπάθησα να σας παρακινήσω και μάλλον τα κατάφερα. Και ελπίζω μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία και να τη συγκεκριμενοποιήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου και στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. We, σας χρειαστεί να ομοιοδοποιήσουμε τις ερωτήσεις αργότερα, αλλά εφόσον έχουμε τώρα μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα σας απαντήσει αμέσως ο υπουργό. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε συνάντηση την περσμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και απλώ θέλω να προσθέσω και τον κύριο Γκοζέ. Φροντίζω να κινούμαστε βήμα-βήμα. Έχουμε ένα σημείο προσανατολισμού τη Προεδρία, το οποίο έγινε ευνοϊκά δεκτό από τις ομάδες στο Κοινοβούλιο. Μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο με συγκεκριμένο νομικό περιεχόμενο σχετικά αφορά το private equity για τις συζητήσεις επόμενης, αυτής της εβδομάδας. Για τις τρίτες χώρες έχουμε ένα άτυπο συμβούλιο τέλος του μηνός για να δούμε εκεί μπορούμε να κάνουμε πρόταση που να την υποστηρίζει το Συμβούλιο. Μακάρι να γίνει αυτή τη βδομάδα, αλλά αν χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη, καλό θα είναι να ξεχωρίσουμε αυτούς τους δύο φακέλους. Σύμφωνα με αυτά που είπατε. Ένα κείμενο για την private equity και οι συνεχίσεις για το διαβατήριο για τις τρίτες χώρες συνεχίζονται. Πρόεδρος, θα αναφέρω τα ονόματα. Philippe, Peter, Dirk, Vicky, uh, Marianne, Marcus, Ferber, Elisa Ferreris, Sven Gold, Sylvie Goulard and Nicholas Shuntis. Uh, Edward, did you... No, and I thought there was another hand down there. If I missed somebody. Μήπως ξέχασα κάποιον. Ο κύριος Κλούτ, Σάντσες Ποσέντο, ο Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Πολύ ευχάριστη η έντονη δράση σας. Έχετε χρόνο να παραμείνετε στην Προεδρία ενώ δεν γίνεται κυβέρνηση στο Βέλγιο. Θετικό αυτό. Τώρα για την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Σωστά είπατε χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία για τις δαπάνες αλλά πρέπει να δούμε και τα έσοδα αναφέρεται την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής. Χρειαζόμαστε και νέους πόρους, προσθέτω. Γιατί ναι, να μειώνουμε το φορολογικό βάρος στο εισόδημα των εργαζομένων, αυτό σημαίνει νέα φορολογικά έσοδα, όπως ο φόρος στις δημοσιονομικές πράξεις. Δεν πολύ αναφέρθηκε σήμερα η φορολογία της ενέργειας ή των πρώτων υλών. Και ήθελα να ξέρω τι πρωτοβουλίες θα πάρετε για να ευνοηθεί μια σύγκληση απόψεων ώστε να υπάρξουν αυτά τα μέτρα και να καταπολεμηθούν οι αντιστάσεις. Γιατί δεν μου επίτροπο σε μέτα πρόβαλε πολλά επιχειρήματα σχετικά με τη φορολόγηση των ε, ε, χρηματοπιστωτικών πράξεων. Μερικά δεν στέκονται από τα επιχειρήματα. Ε, λοιπόν, για, τους νέους, για τα νέα αυτά έσοδα και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι ανάφερε και τη δυνατότητα νέα έσοδα να πάνε κατευθείαν στον προπολογισμό της Ένωσης με αντάλλαγμα μείωση της οικονομικής εισφοράς των κρατών μελών. Ποια είναι η θέση σε αυτού. Και το τελευταίο, η Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ στις πρώτες σελίδες όσο ήταν την Άνοιξη. Κοιτώντας όμως τα νούμερα, βλέπουμε ότι ναι μεν διευκολύνθηκε το άμεσο, η άμεση κατάσταση για την Ελλάδα, πάντως αργά γρήγορα θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος της. Αν όχι για το κεφάλαιο, τουλάχιστον για τους τόκους διαχρονικά. Ποια είναι η θέση σας από αυτού. Έχουμε περίπου 14 ακόμη ομιλητές. Καλό θα ήταν ίσως ε, να ακούμε 3-3 και να απαντά μετά ο υπουργό. ο Πίτερ Σκίνερ. Ευχαριστώ πολύ Σάρον. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σας ε, στο έργο για τις υποδομές. Νομίζω ότι είστε ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς ε, πολιτικούς ε, και βέβαια το δικό μου αφεντικό εξαφανίστηκε για λίγο καιρό με αποτέλεσμα τελικά να μπορέσετε εσείς να συνεισφέρετε τη σοφία σας και το χιούμορ σας και νομίζω ότι έτσι λύθηκε και το αδιέξοδο στη συζητήση σας. Ευχαριστώ λοιπόν για την προσωπική σας συμμετοχή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις συζητήσεις όπως είπατε κι εσείς μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και ΕΠΑ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτιθέλει να κάνει ένα είδος συγκριτικού χάρτη και ενδιαφέρον θα είναι αλλά και πολύπλοκο αυτό το εγχείρημα. Δώδεκα σημεία ε, ήταν ε, σε ένα δικό μου πρόχειρο σχέδιο που έκανα το καλοκαίρι. Βλέπω ότι έχουμε καταφέρει με τα μισά κάτι. Ε, στα 6-7 δεν έχουμε κάνει τίποτα αλλά ούτε και από τη ΣΥΠΑ έχουν γίνει βήματα ότι γίνονται πράγματα και το είπατε και κατά το παρελθόν πολύ σωστά ότι έχουμε και τα περί παγκόσμιας ρύθμισης. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς φαινόμαστε σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ίσως θα έπρεπε και εμείς και εσείς να τα συζητήσουμε ακόμη περισσότερο με τους Αμερικανούς. Αν θέλει κάτι να κάνει η Κομισιόν, αν θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο κάτι, καλό θα ήταν να έρθει κοντά μας, να έρθει στο πλευρό μας και το Συμβούλιο. Να έχουμε το θεσμικό τρίγωνο ενωμένο, γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσουμε τα περιρρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ρέπινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση για τις ε, δοκιμές ε, αντοχής ή κόπωσης, τα λεγόμενα stress tests, τα οποία είδαμε σε διάφορες ε, ευρωπαϊκές τράπεζες να γίνουν τον τελευταίο καιρό και Πράγματι, περισσότερο έγινε αυτό σε ευρωπαϊκέ τράπεζε παρά σε αμερικανικέ. Έχω όμω την εντύπωση ότι πιο πολύ κοιτούμε την ποσότητα εδώ και όχι τόσο την ποιότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών στο λεγόμενο κυρίαρχο χρέος, sovereign debt, έχει κάπως ε, κρυφτεί και στα στοιχεία και στην ε, εξέταση. Αυτή η δοκιμή λοιπόν αντοχής κατά κάποιο τρόπο έγινε έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους υποψηφίους αν θέλετε και λίγο πολύ να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιος θα περάσει και ποιος θα περάσει αυτό το τεστ. Και τελικά ποιες τράπεζες αποτυγχάνουν, αυτές που πάντοτε αποτύγχαναν. Όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες φαίνεται να είναι σώες και αυλαβείς και, και τελικά παρόλα αυτά ακούμε φόβους να εκφράζονται που λένε ότι ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί στο, στη δοκιμή αυτή αντοχής απέναντι στις τράπεζες, να είμαστε ελαστικοί. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να τα επανεξετάσουμε για να δούμε ακριβώς ποια είναι η έκθεση των τραπεζών αυτών σε αυτό το με κυριακό χρέος. Λοιπόν, οικονομική διακυβέρνηση, άμεση φόρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα κτλ. Ας έχουμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Υπουργό. Να απαντήσω πρώτα, λέει ο Υπουργός, σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ για τον κύριο Σκίνερ. Πράγματι θα έχουμε με τον κύριο Μπαρνιέ ε, κάποια συζήτηση για την συνεργασία μας που θα έχουμε έρθει καν του Ατλαντικού. Πρέπει να, πρέπει να καταλάβουμε και πώς έχει πραγματική κατάσταση στη ΣΥΠΑ. Διαβάζω και εγώ τον τύπο, υπάρχουν επίσης και πολλά σημειώματα, ενημερώσεις ε, που λένε ότι θα πρέπει να ψηφιστεί ε, κάποια διάταξη για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στη ΣΥΠΑ κτλ. Τι είδους όμως, τι είδους θα πρέπει να είναι αυτή η χρηματοπιστωτική εποπτεία. Είπαμε ότι θα το συζητήσουμε και με την κυρία Μπόουλς ε, θα μπορούσαμε τον Οκτώβριο να έχουμε μια σχετική συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μπαρνιέ είναι δετεθειμένος ε, να παραστήσει με τέτοια συζήτηση για να δούμε ακριβώς και ποια είναι η πρόοδος ένθεν κακήθνα του Ατλαντικού, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι καταρχάς είναι σημαντικό να εξηγήσουμε κάποιες εξελίξεις. Εξίσου σημαντικό βέβαια είναι και να κάνουμε μια διαφορά Άλλο είναι η ανακοίνωση που λέμε και άλλο είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στον επίσημο, στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ ε, θα το κάνουμε και θα έχουμε και με το Κοινοβούλιο λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νέα έσοδα. Στο τελευταίο ΕΚΟΦΗΝ και το είπα και στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, Είχα λοιπόν τη δυνατότητα να αναφέρω και την τραπεζική εισφορά ως μέσο επίλυσης της κρίσης. Έχουμε εξέλιξη θετική στη συζήτηση και ε, τη φορολόγηση των ε, συναλλαγών. Το δεύτερο θέμα αφορά αρκετά κράτη. Ήδη στο Βέλιο, να αναφέρω το παράδειγμα της χώρας μου, έχουμε ψηφίσει φορολόγηση των τραπεζών και έναν άλλο φόρο, τόμπιν ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τον, Πάντως προχωρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναγνωρίζω και το είπα και στο Στρασβούργο ότι υπάρχουν πολυπλοκότητες. Ό,τι αφορά τη φορολόγηση της ενέργειας, ξέρετε ότι εδώ έχουμε προβλήματα. Τι κάνουμε με την πυρηνική ενέργεια, αφενός, ξέρετε όπως και εγώ, ότι γίνονται κάποιες διαφορετικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις ε, ανάλογα με τις χώρες και ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες. Και αφετέρου το θέμα είναι, είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποια στιγμή μια πρόταση. Αυτό που εγώ είχα προτείνει είναι τουλάχιστον η μιναμαλιστική άποψη να ξαναδούμε την οδηγία για την φορολόγηση της ενέργειας. Μπορούσαμε να δούμε διάφορα σημεία ή να, επανέλθουμε σε, να επανέλθει νέα πρόταση. Δεν έχω μέχρι στιγμής ε, κάποια συγκεκριμένη ένδειξη ότι περιμένουμε ή θα μπορούσαμε να περιμένουμε νέα πρόταση της Κομισιόν. Είπατε επίσης ότι χάρη στο νέο αυτό πόρο θα μπορούσε να μειωθεί η φορολόγια ε, επί της εργασίας και ποια είναι η άποψη της Προεδρίας. Η άμεση εισφορά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, άρα μείωση της, εισφορά, της εισφοράς ε, των κρατών μελών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτού του νέου ίδιου πόρου, έχω ακούσει απόψεις ε, για χρηματοδότηση ε, της προστασίας του περιβάλλοντος. Έχω ακούσει τέτοιες προτάσεις και από πολιτικές ομάδες και από κράτη-μέλη. Άλλοι λένε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη. Ω Υπουργό Οικονομικών ένα πράγμα μπορώ να σας πω πάντως, ότι αν καταφέρουμε τελικά να εισπράττουμε ε, αυτό, μία φορά θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα μπορώ να το κατανέμουμε βέβαια, αλλά όντας 12 χρόνια επικεφαλής ενός Υπουργείου Οικονομικών, με την εμπειρία που έχω αποκομίσει, μπορώ να σας πω ότι μία φορά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, τον πόρο αυτό. Ωραία, μπορούμε να πούμε ότι με το φόρο αυτό μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, να μειώσουμε την εισφορά των κρατών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειώσουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα κτλ. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα κατανεμηθεί ο πόρος αυτός. Δεν θα είναι 100% σε καθένα από αυτούς τους στόχους. Εγώ πρότεινα στο πλαίσιο του ΚΟΦΗ να συζητήσουμε τον νέο αυτό ίδιο πόρο. Δεν μπόρεσε να γίνει κατά το παρελθόν και τώρα μπορεί να γίνει και ελπίζω τους επόμενους μήνες να το καταφέρουμε και να πείσουμε σίγουρα ε, γίνονται ε, κάποιες άλλες προσπάθειες ε, για να έχουμε εξέβρεση πόρων, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια σαφή συζήτηση πάνω σε αυτό. Τώρα στα stress test που είπατε, σε ό,τι αφορά το ECOFIN, Νομίζω ότι είναι πολύ καλή δοκιμή αντοχής που έγινε με την ΕΚΤ και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Χαρακτηρίστηκε από μεγάλη διαφάνεια η άσκηση αυτή σε σύγκριση με αυτό που έγινε σε άλλες χώρες. Πραγματικά ήταν πολύ διαφανής η άσκηση αυτή. Πολύ αποτελεσματικό. Και βέβαια ήταν μια πρώτη απόπειρα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Φυσικά, γιατί όχι. εμείς, ο κ. Μπαρνιέ, εγώ φυσικά και μπορούμε ως μέλη της Επιτροπής να διοργανώνουμε σε τακτά διαστήματα τέτοιου είδους δοκιμές αντοχής. Μία-δυο φορές το χρόνο, για παράδειγμα, θα το δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μπορούμε να κάνουμε τέτοιες δοκιμές, πραγματικές δοκιμές. Τώρα, με την ίδια συλλογιστική, για την ίδια διαφάνεια και αν είναι δυνατόν. Αν μπορεί να γίνει και να το συστήσουμε και σε επίπεδο G20, αν είναι σωστά τα θεμέλια και σωστές οι βάσεις, πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε άλλες χώρες. Είναι οι ίδιες οι παράμετροι, παράδειγμα χάρη, στην ε, Ευρώπη, στην Ασία και στη ΣΥΠΑ. Γιατί οι παράμετροι πρέπει να είναι οι ίδιες και το ίδιο και ο βαθμός διαφάνειας. Αλλά νομίζω ότι ως πρώτη δοκιμή αντοχής ήταν πολύ καλή και αποτελεσματική και διαφανής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον και εγώ θα συνηγορούσα υπέρ της διανέργειας τακτικών τέτοιων δοκιμών αντοχών ίσως να μην περιοριστούν μάλιστα μόνο στις τράπεζες αυτές τις δοκιμές, αλλά και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. γιατί τις τράπεζες είναι χρήσιμο. Γιατί λοιπόν να μην το επεκτείνουμε και σε άλλες χρηματοπιστωτικές ε, εταιρείες, μάλλον όπως παραδείγματος χάρη ασφάλειες. Θα πάω λοιπόν τώρα τη, καταρχήν τη Βίκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, το, για την ε, ολοκλήρωση του θέματος της ε, εποπτείας που ήταν πολύ σημαντικό για τους κινδύνους τους διασυνοριακούς και για τη διοσυνοριακή διαφάνεια για να μπορούν να καθοδηγούνται οι εθνικοί νομοθέτες. Αυτό όσον αφορά την πολιτική ισορροπία. Οι χρηματαγορές είναι ακόμη πολύ ευαίσθητες και φοβάμαι ότι οι αγορές ε, ανησυχούν πάρα πολύ διότι ορισμένες ε, τράπεζες είναι σε πολύ δύσκολη θέση ε, και φοβούνται και το stress test που τους έγινε, δηλαδή τη δοκιμασία αντοχής. Θα πρέπει λοιπόν όπως είπαν ορισμένοι φίλοι μας να εξετάσουμε αυτά που είπαν ορισμένοι πολιτικοί δηλαδή να μιλήσουμε με τον κύριο Τρισέ με τους εμπειρογνώμονες για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα για να ξέρουμε πώς μπορεί κανείς όντως ε, να αντισταθμίσει τον οικονομικό κίνδυνο και επίσης ε, σε μια εφημερίδα διάβασα το Σαββατοκύριακο ότι θα χρειαστούν διεθνή ε, ε, λογιστικά πρότυπα. Πιστεύετε λοιπόν ότι ε, θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να μαγειρεύουν αυτά τα πρότυπα διότι κάποιος μπορεί να πει ότι η δικιά μου αγορά χρειάζεται αυτό ή εκείνο και όσον αφορά το FTT ο, ο Τρισέ την περασμένη εβδομάδα είπε ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο για την Ευρώπη. Πρέπει να τον ακούσουμε. Ευχαριστώ η Άριαν Τάισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω όπως και οι συνάδελφοι να σας συγχαρώ για τα αποτελέσματα που επιτύχατε και έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση όσον αφορά το σχόλιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι θα κοιτάξουμε την συνεκτικότητα ή την απουσία συνεκτικότητας μεταξύ της καταστάσεως των τραπεζών και ε, της προστασίας των ε, ε, Σύβας Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τα σχόλιά σας για την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα και για τα λογιστικά πρότυπα, συμφωνώ με τα σχόλιά σας, δεν θα έπρεπε όμως να εκφράσουμε ε, τις, ε, τις κρίσεις μας σχετικά με τα πρότυπα αυτά, διότι είπαμε ότι χρειάζονται διεθνή λογιστικά πρότυπα για τους ολοκληρωμένους συγκεκριμένους λογαριασμούς για τις εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο. Και τα τελευταία χρόνια ο τρόπος με τον οποίο έγινε ε, το γεγονός αυτό και η αξιολόγηση δημιουργεί διακυμάνσεις και ε, αν ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επενδύσεις όπως το καζίνο ή το λαχείο είναι κακό. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν ενιαία λογιστικά πρότυπα και να να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους καταθέτες. Επίσης, εάν ε, ελέγχεται πώς επενδύει ο κόσμος, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε πολύ κοντά στην κατάσταση του καζίνο και γι' αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ε, τα άτομα για το ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι και επίσης ε, θα, πόσο θα αντιμετωπίσετε μια τέτοια συμπεριφορά. Ευχαριστώ. Καταρχήν χαίρομαι διότι μετά από συζήτηση πέραν του ενός έτους κατάφερα να καταρτιστούν οι κανόνες παιχνιδιού για την ευρωπαϊκή εποπτεία των χρηματαγορών και έχουμε και τα hedge fund αυτή την εβδομάδα θα μας δώσει ε, νέες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τους συμβούλους τις αξιολογήσεις υπάρχουν δηλαδή πολλά ακόμη θέματα που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση των χρηματαγορών και θα ήθελα να, να ξέρω κατά πόσον η η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι έτοιμη να ε, προχωρήσει και να προβεί σε διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Συμβουλίου για να μην χρειαστεί τόσος χρόνος όσο χρειάστηκε για την εποπτεία. Επίσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόκειται να συζητηθεί στην ομάδα εργασίας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού του Προέδρου της Ευρώπης αυτή εποχή ε, η κατάσταση της της, ε, ε, του, της θήκης ε, σταθερότητος και αναπτύξεως γιατί έχω την εντύπωση ότι από το μέσα και με του Μαΐου και μετά δεν μπορούν τα κράτη να καταλήξουν σε συμπεράσματα τουλάχιστον σε ένα επίπεδο το οποίο είναι αναγκαίο για να αξιολογήσουν πώς μπορεί να προωθηθεί το σύμφωνο σταθερότητος και αναπτύξεως. Ε, η Βελγική Προεδρία έχει ακόμη τρεις μήνες καιρό και μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, όσον αφορά τη συζήτηση ε, για τον φόρο των ε, ε, χρηματικών συναλλαγών ή την ανάγκη να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες πρέπει να σας πω ότι με τον κύριο Τρισέ συζητάμε εδώ και 15 χρόνια άρα είναι πολύ έμπειρο στο θέμα αυτό και τώρα είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χρειαζόμαστε βέβαια και εμπειρία εκτός του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά πρέπει στο κάτω-κάτω να βρούμε έναν τρόπο να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Όσον αφορά τον, ε, τη φορολόγηση των ε, χρηματικών ε, ε, συναλλαγών θα πρέπει ε, να οργανωθεί η φορολογία γιατί μπορεί να φορολογήσουμε το νερό θα μου πείτε γιατί όχι ε, όσον αφορά τις χρηματικές ε, συναλλαγές ε, γιατί να μπορούμε να τις φορολογήσουμε ίσως θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε διεθνές επίπεδο αλλά αν φορολογούμε το νερό γιατί όχι τις ε, χρηματικές συναλλαγές Ίσως ε, πρέπει να υπάρξει εμπειρία, θα πρέπει να ακούσουμε πολλές θέσεις, αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Και επειδή η απόφαση στο Βέλγιο έχει ληφθεί εδώ και κάμποσο καιρό, θα πρέπει να, ε, ε, υπάρξει μία γεωγραφική διάσταση σε αυτή τη φορολόγηση. Ε, βεβαίως, ε, χωρίς, ε, αν πούμε ότι χωρίς τις Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποφασίζουμε, χωρίς ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποφασίζουμε ή ε, στην Ευρώπη ή με ορισμένους εταίρους μας διότι για τον, όσον αφορά την, την φορολόγηση των χρηματικών συναλλαγών είδαμε ότι υπήρξε συνεργασία με την Ιαπωνία. Λοιπόν, αν όχι με την Ιαπωνία, με κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν να τι φορολογήσουμε τη στιγμή που φορολογούμε το νερό. Υπάρχει, υπάρχουν τόσοι φόροι υπό τόσε μορφές για τόσα προϊόντα και τόσες υπηρεσίες που γιατί όχι για τι συναλλαγές. Δεν είναι εύκολο ίσω να οργανωθεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Τώρα, Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να αξιολογήσει κανείς, συνεχίζει Ολλανδικά ο κύριος Ρέιντερς. Το είπα αυτό και σχετικά με την απόφαση όσον αφορά τη Βασιλεία διότι πρέπει να υπάρξει μια συνεκτική πολιτική τόσο σε σχέση με την ε, ε, κάλυψη ε, των εθνικών συμφερόντων αλλά ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να εξασκεί και κάποια κριτική και αυτό είναι δύσκολο. Όπως σας είπα λοιπόν τέλος ε, Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε ε, στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ το θέμα αυτό αλλά θα πρέπει να υπάρξει μία επισκόπηση ε, όλων των κανόνων διότι έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις αλλά χρειάζεται και νέος έλεγχος των τραπεζών και τέλος θα χρειαστεί να υπάρξει και μία φορολόγηση τραπεζική για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανείς ε, την οικονομική κρίση. Πώς όμως μπορεί αυτό να ε, ε, συμβιβαστεί με τα καταναλωτικά αγαθά, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διότι και η τραπέζοι ε, τράπεζες εμπλέκονται στην οικονομική πολιτική. Όπως είπα όμως πρέπει να στηρίξουμε και το κράτος διότι εάν καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα παραδείγματο χάρη θα είναι καταστροφικό. Και υπάρχουν και διάφορες απόψεις. Θα προσπαθήσουμε να εξασκήσουμε μία συνεκτική πολιτική και έρχομαι τώρα ή στα πρότυπα της σε ISB. Ε, σας είπα ότι είναι ε, πολύ πιο εύκολο η οι υπουργοί να μιλούν μεταξύ ε, υπουργών οικονομικών και δεν χρειαζόμαστε τόσους εμπειρογνώμονες. Ε, επίσης ε, δεν μπορώ εγώ παραδείγματος χάρη να αναλάβω να κάνω μία συζήτηση σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα. Για μία τέτοια απόφαση θα χρειαζόμαστε μία έκθεση που να έχει καταρτιστεί από εμπειρογνώμονες. Θα πω και στην επόμενη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ θα χρειαστούν εμπειρογνώμονες από πλευράς του Κοινοβουλίου των κρατών μελών και θα να μας πούν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να τα συγκρίνουν με την κατάσταση στις Ηνωμένε να μας πούν πώς μπορούν να επηρεαστούν οι συναλλαγές διότι μία τέτοια σοβαρή τεχνική συζήτηση δεν μπορεί να γίνει στο ΕΚΟΦΗΝ άρθρο προς άρθρο ή να έχουμε τεχνικές συζητήσεις στο ΕΚΟΦΗΝ και ε, τους τελευταίους μήνες άκουσα ότι θα έπρεπε να κάνουμε και κάτι άλλο. Μου ελέγχθη ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε στάση. Θα ήθελα όμως πρώτα πρώτα να υπάρξει μία έκθεση και να ξέρουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ιδίως σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Το είπα και στον κύριο Μπαρνιέ. Χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες οι οποίοι να κάτσουν κάτω και να καταρτήσουν μία έκθεση. Ίσως όχι μία γενική επισκόπηση αλλά σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένα πρότυπα που αναφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης όσον αφορά ε, τα, τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις δεν είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι πρόβλημα των κρατών μελών και ε, ε, παραδείγματος χάρη υπάρχουν ε, ορισμένοι επενδυτές έχουν φορολογικές διευκολύνσεις κατά τρόπον ώστε μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να μπορέσουν να επωφεληθούν. Αλλά αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι είναι και χρήσιμο. Δηλαδή μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα εάν έχει κανείς, αν κάνει κανείς επενδύσεις θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη σε μια κοινή επενδυτική πολιτική. Αλλά αυτή είναι μια πολιτική απόφαση και φαντάζομαι ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να συζητήσουμε π.χ. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έρχομαι τώρα ε, στο τέλος, αλλά μετά από μια επιπλέον ερώτηση. Δηλαδή, θα υπάρξει μία συζήτηση και έχουμε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα χρειαστούμε όπως σας είπα συζητήσεις βασικημένων και περιμένω στις 29 Σεπτεμβρίου για να παραλάβω τις ε, νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το συζητήσουμε με ε, ε, το ΕΚΟΦΗΝ και με την Task Force που θα προτείνει μία λύση για την διακυβέρνηση, την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορέσουμε ε, να ε, ε, το καλύψουμε. Θα συμφωνήσαμε για την εποπτεία, θα συμφωνήσουμε για τις κυρώσει και είμαι αισιόδοξο ότι δεν φτάνει το σύμφωνο σταθερότητο αλλά χρειάζεται και κάποιο σύμφωνο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την κάλυψη των κλιματολογικών αλλαγών και αυτό ε, δεν ε, βασίζεται μόνο εις έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό αλλά χρειάζεται ε, και άλλα στοιχεία δηλαδή να υπάρχουν διάφορες πολιτικές οι οποίες προωθούν την ε, κοινωνική πρόνοια ε, και ούτω καθεξής. Ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τις κυβερνήσεις από ότι είναι ίσως για την Ευρώπη αλλά θα προσπαθήσουμε. Έχουμε τώρα δυσκολίε γιατί έχουμε 8 συναδέλφου που ζήτησαν να μιλήσουν και έχουμε 10 λεπτά μόνο το ρολόι. Μην κάνετε ερώτηση που δεν έχει γίνει ήδη γιατί επαναλαμβάνω έχουμε 8 μιλητέ και 10 λεπτά. Και σα παρακαλώ ή δυνατόν 30 δευτερόλεπτα η ερώτηση γιατί δεν θα υπάρχει χρόνο για απάντηση. Ελίσσα Φεραίρο. Σα ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. για το χρονοδιάγραμμα για το φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και διάφορα τέλη σε βάρος των τραπεζών, διότι πολλές φορές η κάθε χώρα κινείται μόνη της. Μπορεί να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση στο πρόβλημα του να διασωθούν ε, τράπεζες οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο. Επειδή ήμουν εισηγήτρια για το θέμα αυτό, θα είναι θλιβερό να χάσουμε την ευρωπαϊκή μας διάσταση επειδή δεν δίνεται προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Γιατί η κάθε χώρα κοιτάει μόνο τη δική της δουλειά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, καλό όλους τους να κάνουν όλες τις ερωτήσεις και στο τέλος όλες μαζί οι απαντήσεις. Σβέν. Mm, yes, good Στα αγγλικά. Χαίρομαι που ήρθατε πάλι και σήμερα. Μια σύντομη παρατήρηση για την απάντηση που δώσετε στον συνάδελφο Μάρκος Φέρμπερ. Αν δούμε τις αγορές, οι αγορές περιμένουν χρεοκοπία της Ελλάδας. Και το να πούμε ότι μπορεί να συμφωνήσουμε για μερικές κυρώσεις και ήδη συμφωνήσαμε για το εξάμεινο και από εκεί και πέρα κλπ. Αυτό δεν είναι ισχυρή φιλοδοξία σε θέματα συντονισμού οικονομικής πολιτικής και στο ότι δεν υπάρχει οικονομική ενοποίηση στην Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε καταλάβει την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε στην Ευρωζώνη. Η κατάσταση είναι υπερεπίγουσα και χρειαζόμαστε ηγεσία εκ μέρους του Συμβουλίου να κάνει μια θαραλέα πρόταση. Και κάτι τέτοιο δεν ακούστηκε σήμερα. Σιλβί. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ξανά ήρθατε σήμερα εδώ και για όλα σας κάνετε ως τώρα και με μας μαζί. Να αναφερθώ σε ένα θέμα που δεν έχει μεγάλη προτεραιότητα αλλά που είναι πολύ συμβολικό. Είναι η εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης στα διεθνή όργανα. Το ε, χειμώνα ζήσαμε ένα ψυχόδραμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ. Ε, αν είχαμε εκεί μια έδρα, ίσως θα βλέπαμε πιο ευνοϊκά την παρέμβαση του ΔΝΤ. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να σας βοηθήσει αν αποφασίσετε να κινηθείτε στην κατεύθυνση αυτή. Γιατί αυτό το προβλέπουν οι συνθήκες δεν είναι κάτι ξεκρέμαστο, είναι στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπαν, και εγώ θέλω να σταθώ στο τελευταίο σημείο που τυχαίως ρώτησε η προηγούμενη συνάδελφος, σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη συγκυβερνά στην Ελλάδα με το μνημόνιο Υπάρχει απόφαση για έναν ενιαίο χρηματοδοτικό μηχανισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και το ερώτημα είναι, θα συζητήσετε, θα κάνετε και άλλες συμφωνίες, δεν ξέρω τι θα κάνετε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη συνθήκη, άρθρο 218, έχει αποφασιστική γνώμη σε τέτοια περίπτωση. Ποια είναι η δική σας η γνώμη. Θα τα φέρετε αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mr. Klute. Ο κύριος Κλούτ. Ευχαριστώ. Δεν είχε τελειώσει η μετάφραση, γι' αυτό καθυστέρησα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία άλλη και σε ένα άλλο θέμα. Ε, στη Γερμανία παρακολούθησα μία συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση το, της τοπικής αυτοδιοίκησεως των ε, δήμων και κοινοτήτων, η οποία είναι δραματική ε, σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας. Υπάρχουν προσπάθειες ε, μέσω ε, εξοικονομήσεως πόρων να ε, βελτιωθεί αλλά μετά από 15 χρόνια και παρόλη την πολιτική λιτότητα είναι σε χειρότερη κατάσταση και πιο χρεωμένη τουλάχιστον στην περιοχή μου στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία και λένε ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στην κρίση και κληρώνω με αυτό τίθεται το ερώτημα τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουν ε, οι δήμοι και οι κοινότητες να απαλλαγούν από αυτά τα χρέη ε, διότι μέσω αυτών υπάρχει μία πλήρης απόρριψη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο Αντωνίν. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα της υποπτίας θα ασκήσετε τις νέε ευθύνε σας, γιατί είναι σημαντικό θέμα αυτό. Δεύτερον, για την ανάκτηση των πόρων ΩΣΑ, λέω ότι η ανάκτηση είναι σχετικά, η οικονομική ανάπτυξη είναι μέτρια. Ο πρόεδρο Μπαρόσο μίλησε γι' αυτό. Τι σκοπεύει να κάνει το Συμβούλιο σχετικά με αυτό, με την οικονομική ανάπτυξη. Φέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ε, μία ερώτηση σχετικά με την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Δεν ξέρω εάν συμφωνείτε ότι θα μπορεί κανείς να ε, καταπολεμήσει ε, ε, ε, να μπορέσει κανείς να δουλέψει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πρώτο εξάμεινο του 2011 ένα κοινό προϋπολογισμό είναι δυνατόν. Επίσης όσον αφορά τις συνθήκες οι οποίες πρέπει να υπάρξουν για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τα οικονομικά μέτρα. Και τέλος, ο κύριος Καντράουι, θέλω να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ε, όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα διότι πρέπει να υπάρξει μια εταιρική διακυβέρνηση ε, πέραν των οικονομικών μέτρων και πρέπει να ισχύσουν κανόνες παιχνιδιού ενιαίοι πριν από το καλοκαίρι λοιπόν είχε παρουσιαστεί μια πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να ξέρω εάν εσείς θεωρείτε ότι η συζήτηση αυτή είναι σωστή, αν θα συζητηθεί στο Συμβούλιο και αν ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηροί κανόνες στο μέλλον κατά τρόπον ώστε ολόκληρο η Ευρώπη να ε, διεκπεραιώνει με το τρίτο τρόπο τους ε, ελέγχους κινδύνων με συγχωρείτε διότι υπερβήκαμε λίγο το χρόνο μας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ε, μία φορολόγηση των τραπεζών και θα συμφωνήσουμε ε, σε ένα κείμενο, θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε στο κείμενο αυτό στο τέλος του μηνός. Διότι στο Βέλγιο προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρίς όμως να ισχύσει σε άλλη χώρα και ίσως εφέτος μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω διότι αυτό ήταν το 2001 στο Βέλγιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα επ' αυτού αλλά θα προσπαθήσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Δεν είμαι αντίθετο στη συζήτηση. Πρέπει να σας πω δεν καταλαβαίνω τι είπατε σχετικά με την Ελλάδα διότι στην Ελλάδα η κατάσταση είναι καταφανής και συμφωνή συμφώνησαν όλα τα κράτη-μέρη. Ε, και ορισμένοι όπως ο Ζων Κρότρισε και η Γερμανία ε, συμφώνησαν για την Ελλάδα. Ε, συμφωνήσαμε όλοι και μπορέσαμε να βοηθήσουμε. Ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό στο τελευταίο Συμβούλιο και η εξέλιξη στην Ελλάδα είναι πολύ καλή και συνάδει με τις απαιτήσει της Κεντρικής Τραπέζης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου. Ε, εάν εσείς θέλετε κάτι παραπάνω, ίσως θα πρέπει να συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο στη Γερμανία. Διότι ε, αν θέλετε να πείσετε τον Bundestag ή τον Bundesrat να κάνουν περισσότερα για την Ελλάδα, είναι δικό σας θέμα. Εμείς στο Συμβούλιο συμφωνήσαμε να βοηθήσουμε και συμφώνησε και η Γερμανία και έκτοτε είδαμε μία πολύ καλή εξέλιξη η οποία συμφώνεται με τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων και ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όλοι όλοι είχαν συμφωνήσει να βοηθήσουν την Ελλάδα πριν τους Σλοβάκους ε, που δεν το δέχονται και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να κάνουν και κάτι παραπάνω. Ως προς την κυρία Γκουλάς θα ήθελα να της πω ότι ε, θα θέλαμε να προχωρήσουμε αλλά πρέπει να ε, πείσουμε τους πάντες τις μικρές, τις μεγαλύτερες και τις πιο μεγάλες χώρες της Ευρώπης ότι πρέπει να συμπτυχθούν να συνενωθούν που είναι δύσκολο αλλά αυτό που έγινε στην Κοπεχάγη είναι ίσως ένα πρώτο βήμα διότι αν πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος των εργασιών βρισκόμαστε εκτός συζητήσεως και καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα δεν το στο τέλος των συζητήσεων στην Κοπεχάγη. Ε, βέβαια ήθελα να σας πω ότι ο Ρι Σπακ είχε πει ότι όλα τα κράτη της Ευρώπης είναι μικρά αλλά ορισμένοι δεν το ξέρουν ακόμη. Ίσως επ' αυτού πρέπει να γίνει κάποια προεργασία αλλά δεν θέλω να προχωρήσω περαιτέρω απλώς θα τα έκανα μια ιστορική υπενθύμηση επί του θέματος. Όσον αφορά την εξέλιξη των ε, ελλημάτων ε, στα διάφορα κράτη, το ΕΚΟΦΗΝ απευθύνεται στα κράτη και γνωρίζοντας το Βέλγιο καλά, πρέπει να σας πω είναι πολύ δύσκολο να πείσει κανείς τα κράτη να οργανωθούν με την τοπική αυτοδιοίκησή τους. Σκεφτείτε λοιπόν να συζητάμε τη συζήτηση ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ολόκληρης Ευρώπης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περίπλοκο και γι' αυτό στις συστάσεις τις οποίες μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διατυπώνουμε για τα προγράμματα σταθερότητα θα πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης να δώσουμε καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές αλλά είναι βασικά ε, η ευθύνη των εθνικών αρχών για να μην σας πω των περιφερειακών αρχών επί του θέματος. Όσον αφορά την αύξηση των επενδύσεων στην ε, Ευρώπη. Βέβαια, ε, σας είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη ε, διορατική πολιτική και να υπάρχουν κοινοί κανόνες για τις τράπεζες, για τα μπόνους, για το χρηματοοικονομικό τομέα. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Ξεκινήσαμε την εποπτεία. Έχουμε προτάσεις και ιδέες για διάφορα θέματα για διάφορου τομεί, αλλά είναι μακρύς ο δρόμος για να μπορέσουμε να οργανωθούμε και είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε τις επόμενε συζητήσει στο G20 για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε ορισμένους κανόνε όσον αφορά την πολιτική ε, της ε, ε, ε, των αμοιβών. Όσον αφορά την διακυβέρνηση, τι συζητήθηκε και στους τριμερείς διαλόγους. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιωθεί στην Ευρώπη η οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι κατά καιρού θα πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των Ευρωβουλευτών και των ομολόγων τους των Εθνικών Κοινοβουλίων και μέσω των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνεται το ίδιο πράγμα και στα εθνικά κοινοβούλια διότι χωρίς να θέλω να αναφέρω καμία συγκεκριμένη χώρα καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο έχουμε διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη αλλά και τελείως διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς μεταξύ των ευρωπαϊκών θέσεων και των εθνικών θέσεων και το λέω με μεγάλη άνεση γιατί θα μου πείτε ότι ε, χειρότερα συμπεριφέρονται οι κυβερνήσεις αλλά ε, αν θέλετε να υπάρχει μία προεδρία ε, τώρα η Βέλγικη μετά η Ουγγρική και έχει ο Θεός για να βελτιώσει την διακυβέρνηση θα πρέπει να συντονιστούν οι θέσεις των Ευρωβουλευτών και των Εθνικών Βουλευτών σε κάθε χώρα και σε κάθε πολιτική ομάδα. Εάν υπήρχαν αυτές οι θέσεις τουλάχιστον ήταν πιο εύκολα να πείσουμε τους συναδέλφους γύρω από το τραπέζι αλλά τα προβλήματα είναι ακόμη πιο σοβαρά στο επίπεδο του Συμβουλίου και ευχαριστώ όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επίτευξη Ευρωπαϊκών Συμφωνιών προς ε, άτος. Αλλά όπως σας είπα τις επόμενες ημέρες η συζήτηση αυτή θα γίνει και ο κύριος Γκοζές το ξέρει για μια πολύ σημαντική οδηγία. Ευχαριστώ. για την εταιρική διακυβέρνηση θα δούμε αν γίνεται να έχουμε πρόοδο. Θα το δούμε. Αλλά προς το παλόν ας οργανώσουμε μια καλύτερη διακυβέρνηση. Όπως είπα πριν ε, από λίγα λεπτά για την Ευρώπη και το Συμβούλιο για τους διάφορους εταίρους. Ε, οικονομική διακυβέρνηση κυρίως. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, το συζητάμε στο ΕΚΟΦΗΝ, αλλά υπάρχουν ε, και σε άλλου σχηματισμού του Συμβουλίου συζητήσει από αυτού. Εγώ είμαι ανοιχτό για συμπερίληψη του θέματο στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη όσον αφορά τι επιχειρήσει, σε ό,τι αφορά τι εταιρείε. Άλλο για την ανταγωνιστικότητα και την εσωτερική αγορά. Πάντω, εγώ είμαι ανοιχτό. Θα προσπαθήσω κάτι να οργανώσω. Η πρόεδρο. Σύντομα, λοιπόν, έρχεται και αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή μας θα συναντηθεί με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Μάρτιο θα θέσουμε και το ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκό εξάμεινο, στο πλαίσιο των συζητήσεών μας. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε και να νιώθετε ότι και εμείς κάνουμε τη δική μας ε, δουλειά εδώ. Κάποιοι λένε, μα πώς μπορούμε να γεμίζουμε το χρόνο μας εδώ στην Επιτροπή την Οικονομική. Βλέπετε όμως ότι μπορούμε να μείνουμε ώρες και ώρες να συζητούμε αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και σίγουρα θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Don't go. We've got to do the report back on... Φύγετε γιατί έχουμε την έκθεση για την εποπτεία. Okay, if we could settle down everybody. Παρακαλώ καθίστε. Σημείο... Όχι το 4. Έχετε μία... Όχι δεν είναι το 4. Είναι τα απορίσματα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για την ε, το πακέτο χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Όπως ξέρετε είχαμε ένα τελικό τριμερή διάλογο, μια προσωρινή συμφωνία. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο και Συγγετή ε, Γκαρσία Μαργκάγιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λέει γραμματέα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι γιατί είναι πολλοί συγητές. Θέλω πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Υπουργό που μόλις έφυγε, προς την Κομισιόν, προς τους ηγητές, προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, ε, το Προεδρείο γενικώ, αλλά και τη Γραμματεία που μας βοήθησε. Νομίζω ότι ουσιαστικά κάναμε καλή δουλειά σε αυτή τη συμφωνία με το Συμβούλιο. Δύσκολο ήταν το έργο μας. Για πρώτη φορά έπρεπε να φτάσουμε έξι εισηγητέ με έξι σκιώδεις και συντονιστές, πολιτικές ομάδες κτλ. Έπρεπε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και τα καταφέραμε. Φτάσαμε σε συμφωνία. Παρότι φαινόταν να είναι ένα, το δωμάτιο των αδελφών Μάρξ το, η αίθουσα στην οποία συναντιόμαστε ορισμένε φορέ. Οκτώ μήνε ε, λοιπόν ε, κράτησε όλη αυτή η συζήτηση και είχαμε ευχάριστε εκπλήξει, νέου συνασπισμού, νέε συμμαχίε μεταξύ πολιτικών ομάδων που μέχρι πρότινος φαινόταν να είναι σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και μάλιστα μέχρι και οι Βρετανοί συντηρητικοί ζήτησαν περισσότερες εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έκαναν και έπλεξαν και το εγκόμιο που είναι πραγματικά πρωτάκουστο. Τέλος πάντων, είχαμε κάποιους κινδύνους να πείσουμε. Η κρίση θα μπορούσε να είχε δύο διεξόδους αντιφατικές και διαφορετικές μεταξύ τους. Την επανακρατικοποίηση των οικονομικών πολιτικών όπως έγινε στην αρχή της ε, κρίσης ή περισσότερη Ευρώπη. Αυτές ήταν οι δύο επιλογές όπως έλεγαν οι ε, δύο εκθέσεις Λαροζιέρ και Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της επανακρατικοποίησης φαινόταν ότι θα υλοποιηθεί αυτό. Ήταν σαν ε, ρώσικες κούκλες. Κάθε κούκλα που ανακαλύπταμε ήταν ε, όλο και πιο μικρή και όλο και πιο ασήμαντη. Η έκθεση Λαροσχέρ ε, ε, υποτιμήθηκε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο υποτίμησε την έκθεση της Κομισιόν. Και τελικά ακούσαμε ότι έπρεπε στην ομάδα Λαροσχέρ ε, αυτή η όθηση και αυτή η ορμή που υπήρχε να ανακτηθεί με κάποιο τρόπο και αυτό τελικά έγινε. Αυτό το οποίο καταφέραμε ήταν να ψηφίσει το Κοινοβούλιο στις 7 Ιουλίου κάποιες τροπολογίες με μαζική υποστήριξη, τροπολογίες που ήταν αντίθετες σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις ε, του Σουηδικού Συμβιβασμού. Αλλά αντί να έχουμε με τοπική σύγκρουση, τελικά καταφέραμε να έχουμε μια αίσια έκβαση, ένα αίσιο πέρας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ε, βασικές πτυχές της έκθεσης και σε κάθε μέλος επιτροπής ε, έχω να δώσω μια έκθεση η οποία έχει δύο στήλες. Ε, στην αριστερή στήλη έχουμε τη συμφωνία του Συμβουλίου που είμαστε αντίθετοι και η δεύτερη στήλη, η δεξιά, είναι η τελική συμφωνία με άλλους χαρακτήρες για να δούμε ποια είναι και η προστιθέμενη αξία και η εισφορά του κοινοβουλίου που είναι σημαντική. Να κάνω τέσσερις αποχρώσεις να δώσω. Σε ό,τι αφορά ε, τις, τις ε, ελεγκτικές αρχές ε, της Ευρωπαϊκής το καταφέραμε ενώ ήταν, υπήρξαν αντιδράσεις. Θέλουμε επίσης και καταφέραμε να έχουμε αρχές με ισχύ. Αδόλφο, σε παρακαλώ. Αρχές λοιπόν οι οποίες θα μπορούν να προτείνουν ε, κάποιους κανόνες ανάπτυξης και εκτέλεσης ώστε όλοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να υποβάλλονται, να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες σε όλη την κοινοτική επικράτεια και υπάρχουν επίσης και προσανατολισμοί, κατευθύνσεις και συστάσεις όταν δεν υπήρχε νομικός κανόνας συγκεκριμένος. Οι αρχές αυτές λοιπόν θα μπορούν να διασφαλίσουν την υλοποίηση των κανόνων που προτείνουν και αναπτύσσουν. αν υπάρχει αδράνεια των ε, εθνικών ε, ελεγκτών ή αν δεν υπακούει εθνικός ελεγκτής ε, στις αποφάσεις ερικής αρχής, θα πρέπει τελικά να υποκληθεί στις, στους κανόνες αυτούς. Η συμφωνία του Συμβουλίου, κατά την άποψή μου, στρεφόταν ιδιαίτερα προς τις αρχές, ενώ εμείς αποφασίσαμε να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των χρηστών, των τραπεζών, με τη δυνατότητα απαγόρευσης ορισμένων τοξικών συμφωνιών, με την ενσωμάτωση της μικρομεσαίας επιχείρησης στους συμβουλευτικούς φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε θέματα χρηματοπιστωτικής πολιτικής και λάβαμε επίσης υπόψη κάτι που το Συμβούλιο δεν είχε λάβει υπόψη στην αρχική του έκθεση ούτε και Επιτροπή η Ευρωπαϊκή. Δηλαδή του συστημικού κινδύνου. Εμείς είπαμε ότι ένα μείζον ζήτημα ε, στο πλαίσιο αυτής της κρίσης ήταν να επιληθεί η κατάσταση κατά την οποία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πολύ μεγάλα για να χρεοκοπήσουν όταν ε, ουσιαστικά καταπατούν τη βασική αρχή, δηλαδή όταν κάποιος ε, σε σχέση με τη χρεοκοπία. Δεν μπορούσαν δηλαδή να χρεοκοπήσουν παρότι καταπατούσαν τους ε, βασικούς κανόνες. Αυτός λοιπόν ήταν ο συστημικός ε, κίνδυνος. Θα έχουμε αυτές τις ε, δοκιμές αντοχής που για πρώτη φορά θα είναι ομοιογενείς και αξιόπιστες και θα παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενισχυμένη εποπτεία για φορείς και ιδρύματα που δίνουν κάποια δείγματα κόπωσης ή πιθανής χρεοκοπίας πτώχευσης. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προχρηματοδοτούν ε, το, τα, τα εναρμονισμένα ταμεία και τα άλλα ταμεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να ε, υπάρξουν οι απαραίτητες πληρωμές όταν χρειαστεί. Άρα οι ελεγκτικές αρχές που είναι ισχυρές και που υποβάλλονται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου, άρθρο 7 λοιπά, δείχνουν το ρόλο που θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη των ρυθμιστικών κανόνων και των κανόνων ανάπτυξης. Καταφέραμε έτσι να λύσουμε ένα πρόβλημα που είχαμε αντιμετωπίσει ήδη από, από το Λαμφαλουσί. θα υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτές οι νέες αρχές με έναν καινοτόμο και θα έλεγα και πολύ πιο απαιτητικό τρόπο σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει στο νομισματικό διάλογο με τον πρώτος κεντρικής τράπεζας. Θα πρέπει να γίνεται μια προκατακτική γραπτή έκθεση, μετά έκθεση στην οποία θα αναφέρουμε τα ζητήματα που μα ενδιαφέρουν, τι δεν έγινε, ποιε είναι οι διεθνεί συμφωνίες, ποιε χώρες έχουν εκπληρώσει τι ε, υποχρεώσει, ποιε όχι κτλ. Και έτσι λύνεται αυτό το πολύ λεπτό θέμα του accountability, της ε, υποχρέωσης λογοδοσίας. Ολοκληρώνοντας να πω ότι κάναμε καλή δουλειά κατά την άποψή μου, φέραμε σε πέρα στην αποστολή που μας ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η δουλειά της γραμματείας και πιστεύω ότι και αυτός ο τριμερής διάλογος είναι το πρώτο βήμα ε, προς μια κατεύθυνση για την αποτοπιστωτική εποπτεία με ευρωπαϊκή εστίαση και επίκεντρο και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Κάτι το οποίο ζητούσαν και οι Ευρωπαίοι πολίτε που μα έφεραν με την ψήφο του στα έδρανα αυτά. Ολοκληρώνω εδώ και ελπίζω ότι και με την έκθεσή μου, με αυτέ τι στήλε που τι έχετε, έχετε αυτό το έγγραφο, μπορείτε να το μελετήσετε στον υπολογιστή σα και ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι πραγματικά ήταν καλή δουλειά και αξίζει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Thank you Ευχαριστώ. Τώρα... Ε, θα περάσουμε στην ε, αρχή ε, των αγο... Ε, ε, ρυθμίσεως των αγορών. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν και όλα τα ευχαριστώ, αλλά θέλω να τονίσω δύο επιτεύγματα. Καταρχήν ότι Έχουμε αυξήσει τις αρμοδιότητές μας όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και θα πρέπει να επιμείνουμε ασχέτως εάν χρησιμοποιηθούν ή όχι αυτές οι αρμοδιότητες και δεύτερον θα ήθελα να εμποδίσουμε την εμπορία ορισμένων προϊόντων διότι ακόμη και μετά την ε, ε, ψηφοφορία θα έχουμε διάφορες δυνατότητες διότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματά της μιλούσαν για προσωπικό 100 ατόμων για το νέο θεσμικό όργανο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μέγεθος το οποίο πρέπει να επιζητήσουμε διότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τους αναγκαίους πόρους γιατί τουλάχιστον στη Γερμανία έχουμε διαπιστώσει ότι δεν αξίζει τον κόπο να έχουμε θεσμικά όργανα τα οποία δεν έχουν σωστό προσωπικό, δεν έχουν επαρκές προσωπικό και σαν κοινοβούλιο θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, δηλαδή πώς και ποιος θα επανδρώνει τι. Επίσης, ε, εις ε, την ε, οδηγία για την ε, διαφάνεια είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμευτεί να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση μέχρι ε, το φθινόπωρο του επομένου έτους. Οπότε εμείς σαν Κοινοβούλιο πρέπει να δούμε τι θέλουμε, να καταρτήσουμε μια έκθεση για να συζητήσουμε ποια είναι η κατάσταση. Και τέλος, Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να προετοιμαστούμε και να προετοιμάσουμε την ε, συνεισφορά μας ε, ε, στο ποιος θα αναλάβει την, να είναι επικεφαλής του θεσμικού αυτού οργάνωση. Όχι αυτό το οποίο αναφέρεται η Σιλβή, αλλά στην ίσας, διότι εάν υπάρχουν αυτές οι οργανώσεις και γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ε, ε, απολογούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αυτή την Επιτροπή, ε, τότε θα έχουμε καλύψει αυτό για το οποίο μας έχουν ψηφίσει. Σαν συντονιστές λοιπόν, αφού επιτύχουμε το συμβασμό με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπάρξει μία υποδομή της αγοράς υπό ε, ε, ε, ε, υπό εποπτεία κατά τρόπον ώστε να μην επανέλθουμε στην ίδια συζήτηση όταν θα μιλήσουμε για τα χρηματοοικονομικά παράγωγο διότι θα πρέπει να κατανοήσουμε τις ε, ε, αυτά τα θεσμικά πλαίσια τα οποία καταρτίζουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και θα το ξαναδούμε διότι έχουμε από κοινού ψηφίσει για αυτές τις αλλαγές. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Πίτερ σχετικά με τις επαγγελματικές ασφαλίσεις. Ευχαριστώ. Ε, είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι Δεν έχει σημασία πάντοτε πόσο μεγάλο είναι το σκυλί που παλεύει, αλλά πόσο θέλει να παλέψει ένα σκυλί. Αυτό λοιπόν που ε, λέχθη προηγουμένως για το μέγεθος των οργανισμών ε, αυτών είναι ε, κάτι το οποίο συζητήθηκε αρχικά εις τις διαπραγματεύσεις που εγκαταλείψαμε και πρέπει να ξανασυζητήσουμε διότι τα 90 ή 100 άτομα να οργάνωση οργάνωση δεν ε, θα καταρρύψει ή θα διακενδυνεύσει διάφορα κράτη διότι ε, αν δείτε ε, πόσο περίπλοκα είναι τα συστήματα στις Ηνωμένε Πολιτείε, θα αντιληφθείτε ότι έχουν να ανταποκριθούν σε ένα πολύ σοβαρό έργο. Στις αρχές του 2011 θα έχουμε συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να απαντούμε σε διάφορα ερωτήματα και να ε, κινητοποιήσουμε τα άτομα που θα πρέπει να αποφασίσουν για ε, να αντισταθμίσουν το συστηματικό κείμενο, κίνδυνο ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί εάν ε, προκύψει μία τέτοια οικονομική η οικονομική κρίση. Να μην έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τους υπουργούς με τις πιτζάμες τους να πρέπει να προσπαθήσουν μεταξύ τους να συζητήσουν πώς θα αντεπεξέλθουν. Θα πρέπει να έχουμε μια εποπτική αρχή η οποία θα εμπλέκεται και ε, γι' αυτό χρειάζεται μια κοινή επιτροπή την οποία ενετόπισε το Κοινοβούλιο όπου θα πρέπει να έρχονται οι μακροοικονομικές πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Κοινοβούλιο, όπου θα συζητάμε ε, την κατάσταση ε, των διαφόρων εποπτικών αρχών ε, μέρα με την ημέρα και που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και δεύτερον θα ήθελα να πω ότι οι ασφάλειες δεν μοιάζουν με τις τράπεζες και ε, το πρώτο πράγμα το οποίο είχαμε γράψει είναι τι θα επηρεάσει την, ε, τις τράπεζες. Και μετά προχωρήσαμε στη ρύθμιση ε, των ασφαλιών. Τώρα όμως πρέπει να, να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για μακροπρόθεσμους οργανισμούς και θα πρέπει με την ε, Βασιλεία 2 που ασχολείται με την ε, επάρκεια ε, των κεφαλαίων να ξαναεξετάσουμε τα θέματα αυτά. Πέραν αυτού όμως ε, θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να επιλύουμε τις διαφορές διότι αυτό δεν υπήρχε στην Βασιλεία 2 και θα πρέπει να βρούμε διαδικασίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις μας και να υπάρχει και μία δυνατότητα ε, νομικής ή δικαστικής αποκαταστάσεως. Και είναι βασικό διότι πρέπει οι άλλοι να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε σοβαροί όταν νομοθετούμε στην Ευρώπη και διαφορετικά θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε τη Βασιλεία 2 διότι ε, θα πρέπει να βρούμε ένα ψήφισμα το οποίο θα επιλύσει την κατάσταση που δημιουργείται στην Ευρώπη και αν δεν βρεθεί μια λύση γρήγορα πρέπει εμείς να πιέσουμε τα πράγματα. Τέλος πιστεύω ότι οι οργανισμοί θα εργαστούν σωστά. Ε, βλέπουμε ε, πώς επιλέγουν τα, τα πράγματα. Και τέλος πιστεύω ότι οι τράπεζες είναι διαφορετικές. Έχουμε λίγο χρόνο για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει ε, και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι και πιστεύω ότι η ομάδα του Κοινοβουλίου έχει εργαστεί πολύ καλά. Προσβλέπω στους συναδέλφους με τους οποίους έχω συνεργαστεί και τους ευχαριστώ και είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πίτερ ή Σιλβί. Πολύ σύντομα. Ο καλύτερο τρόπο για να δείξουμε ότι συμφωνούμε είναι να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Μην παρατηρήσει Γιατί δώσαμε μάχη για την προστασία του SAB από την Κεντρική Τράπεζα. Διότι θέλουμε να έχουμε μία ανεξάρτητη αρχή που να μπορεί να είναι αντίβαρο στο Συμβούλιο που ζήτησε τη δυνατότητα να καλεί το χαρακτήρα του επίγοντος. Ένα διάλογο που απέναντί του έχει το Συμβούλιο, όπως το ξέρουμε. Δεύτερη παρατήρηση. Καταλήξαμε στο αποτέλεσμα αυτό, διότι υπήρξε η συμφωνία μεταξύ του εισηγητή, αλλά και μεταξύ των ομάδων. Και οι θέσεις μας ήταν φιλόδοξες. Και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτό το πνεύμα όσο γίνεται. Έτσι, για να μείνω στο SIB, πετύχαμε επίσης άνοιγμα των αποφασιστικών οργάνων για τα οποία το Συμβούλιο στην αρχή δεν συμφωνούσε. Προτιμούσε την ενδογαμία των κεντρικών τραπεζών. Θα δώσουμε και άλλες μάχες στο μέλλον, το είπε και ο ΣΒΕΜ. Έχουμε μια δήλωση των συντονιστών, όπου λέμε ότι ό,τι δεν πετύχαμε τώρα, όσον αφορά την εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι αξιολογητικοί οργανισμοί, δομή της αγοράς κλπ, να τα πετύχουμε με τομεακά κείμενα, με επιμέρους κείμενα. Ας συνεργαστούμε όλοι μαζί, οι συγητές, προκειμένου να υπάρχει μια θέση μη ανακολουθίας του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και πάρει όλους και ιδιαίτερα τη Γραμματεία που βοήθησε με μεγάλη προσπάθεια. Ο Ρεμό είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. αρχίσουμε στην, αρχίσουμε στην οδηγία Omnibus 1 που τροποδολογεί όλες τις άλλες οδηγίες. Βέβαια δεν είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο στην Επιτροπή μας σε σχέση με άλλα θέματα, αλλά μην υποτιμούμε την τεράστια δουλειά που έχει μπει στο Omnibus 1 με στόχο το Omnibus 2 αργότερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για τα λόγια σας και για τη συνεργασία που είχαμε και με τους ε, υπόλοιπους ε, συντρόφους ε, εισηγητές, συντάξεις τροπολογικών που είχαμε λοιπόν για να φέρουμε σε πέρα σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι θετικό ο απολογισμό. Στόχο μα ήταν να ενσωματώσουμε στο σύνολο των 11 τομεακών οδηγιών τις μεταρρυθμίσεις που θεσπίζουν νέε ρυθμιστικέ αρχές. Αυτό ουσιαστικά ήταν να περάσουμε από τη διακυβερνητική λογική στο πλαίσιο της εποπτείας σε μια λογική βασισμένη σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ευρωπαϊκών αρχών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό κάναμε και για τις 11 οδηγίες. Ενισχύσαμε την τομεακή συνεργασία, θορίσαμε όρους για μεσολάβηση ε, και ε, προσθέσαμε και κάποια θέματα σε ό,τι αφορά δηλαδή την εκπαίδευση. Θεσπίσαμε επίσης ε, τις νέες αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία της Λισαβόνας που γνωρίζουμε ότι τροποποιούσε όλα τα περί διαδικασίας επιτροπής. Έχουμε τώρα τις ε, κατεξουσιοδότηση ε, πράξη ε, και τις διαδικασίες υλοποίησης, διαδικασίες εκτέλεσης. Στόχος ήταν να έχουμε και τη τεχνική συνεισφορά στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας και νομίζω ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη λύση. Θέλαμε επίσης ε, η εφαρμογή της νέας ρύθμισης να είναι αποτελεσματική. Έχουμε λοιπόν τους ε, πίνακες συσχέτιση στην οδηγία. Ήταν φιλοδοξία του Κοινοβουλίου σε οριζόντιο επίπεδο, αυξήσαμε τη διαφάνεια, θα έχουμε μια κοινή νοοτροπία, κοινή κουλτούρα για την ενημέρωση Θέλουμε επίσης να προετοιμάσουμε τις οικονομικές αρχές για τα σχέδια ανάκτησης και επίλυσης με βάση τα μέτρα και τις απαραίτητες συμφωνίες και υπάρχει και μια πτυχή που ακόμη δεν έχουμε καταφέρει την νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή τις καταχώρα ρυθμίσεις. Πάντως αυτό που καταφέραμε είναι να υπάρχει μια ανακοίνωση, μια ανακοίνωση που θα λαμβάνεται υπόψη και σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για διαφάνεια κατά το επόμενο έτος. Για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερε είναι θετικό βήμα. Φυσικά, κυρία Πρόεδρε, δεν εξαντλούνται εδώ οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες αρχές, αλλά αυτό θα είναι αποτέλεσμα, από αντικείμενο μιας ακόμη σε βάθος εξέτασης και μεταρρύθμισης και θα δούμε και σε αυτό το χρόνο ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, and, and I would add... Ευχαριστώ πολύ να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Αντωνιέ για, για την προσθήκη πινάκων και των κανόνων για τις ε, πράξεις εκχώρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το Κοινοβούλιο σε όλες, από όλες τις ομάδες όσον αφορά την διοργανική συμφωνία. Χαίρομαι για το ότι η Επιτροπή μας υπήρξε πρωτοπόρα στο θέμα αυτό. Οι περισσότερες ομάδες στην Επιτροπή είπαν ότι υποστηρίζουν τον συμβιβασμό. Υπάρχει κανείς που θα ήθελε να πει κάτι αυτή τη στιγμή που να θέλει κάποια διευκρίνηση. Όχι. Το σχέδιο έκθεσης έχει υποβληθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση την Τρίτη, ψηφοφορία την Τετάρτη. Δεν θα έχουμε πλήρη συζήτηση την Τρίτη, γιατί ήδη έχει γίνει συζήτηση. Θα γίνει συζήτηση ή όχι. Την τρίτη τίποτα. Πριν την ψηφοφορία την Τετάρτη θα δοθεί η ευκαιρία στους εισηγητές να πούνε δυο λόγια. Όχι δεύτερη συζήτηση. Δυστυχώς το προσπαθήσαμε, αλλά δεν μας το επέτρεψαν. Και τώρα ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το σημείο θέμα ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα dark pools, διαφανείς δεξαμενές και το σχέδιο της συζήτηση του σχέδιου έκθεσης K. Swinburne. K. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια ως τώρα από τους σκιώδεις και τους βοηθούς και τους πολιτικούς συμβούλους για να φτάσουμε ως εδώ, στην έκθεση αυτή ιδίας πρωτοβουλίας. Ξεκινήσαμε με, δύο, με δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το πρώτο, η οδηγία MIFID πέτυχε αυτό που ήθελε να πετύχει. Και δεύτερον, πρέπει να τροπολογηθεί για να αντιμετωπίσει διερθρωτικές μεταβολές στις χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Στο πρώτο ερώτημα, καταλήξαμε στο ότι ήταν επιτυχής η MIFID στο στόχο της. Έχουμε ανταγωνισμό για την εκτέλεση πράξεων αύξηση των επιλογών για τον επενδυτή, μείωση του κόστους και η διαδικασία δημόρφωσης των τιμών επίσης βοηθήθηκε. Βόηθησε την ενιαία αγορά, αλλά πρέπει να υπάρχει προστασία επαρκής. Το δεύτερο όρτημα λοιπόν, η διαφάνεια στις διαδικασίες πριν και μετά τις πράξεις είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι και υπάρχουν ορισμοί, εξαιρέσεις κλπ. που να ισχύουν σωστά. Και υπάρχουν και ορισμένε προτάσει στην έκθεση. Παράλληλα με την εφαρμογή τη MIFID, η διάρθρωση των αγορών μετοχών στην Ευρώπη άλλαξε. Τώρα έχουμε μεγάλη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι τεχνολογίες δημιουργούν νέες εμπορικές στρατηγικές μεγάλης ταχύτητας, collocation, χρήση αλγορίθμων. Το κόστο και το όφελος όλων αυτών έχουν αναλυθεί Χρειάζονται όμως πάρα πολλά στοιχεία για να καταλάβουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην αγορά και πώς συμβάλλουν στην ρευστότητα και γενικά στην καλή λειτουργία της αγοράς. Ας χρησιμοποιούμε την ευκαιρία να θεωρήσουμε τα βασικά στοιχεία της ΜΥΦΙΤ και τον στόχο της, να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις, για να έχουμε το ενίο της αγοράς και τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια και οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να εξυπηρετούν τις βιομηχανίες και τους επενδυτές. Η έκθεση λοιπόν κατέληξε ότι η ποιότητα των στοιχείων της αγοράς δεν είναι επαρκής. Και πιο συγκεκριμένα, η αναφορά των στοιχείων αυτών για τον πράξενο OTC πρέπει να βελτιωθεί και να προτυποποιηθεί για να έχουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα πληροφοριών και για αυτούς που παίρνουν μέρος στην αγορά, δηλαδή τους χρηματιστές και τους επενδυτές και τους ρυθμιστές. Όταν ξεκινήσαμε την έρευνα τον Απρίλιο, είδαμε ότι η αγορά λειτουργούσε σωστά όσον αφορά την εφαρμογή της MIFID. περιμένουμε λοιπόν να έχουμε αύξηση του ποσοστού από το OTC στις πολυμερείς πλατφόρμες εφόσον είχε υπάρξει ανταγωνισμός. Αυτό όμως δεν συνέβη. Γι' αυτό αρχίζαμε να παίρνουμε στοιχεία από όπου μπορούσαμε, γιατί είναι υπέρ των πράξεων το OTC και γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ε, κινούνται στα λεγόμενα δίκτυα διαφανείς δεξαμενές. Ορισμένοι επενδυτέ προτιμούν να λειτουργούν μέσα διαφανεί αυτέ δεξαμενέ, ιδιαίτερα τα OTC, γιατί θεωρούν ότι διάφορα trade venues δεν τους εξασφαλίζουν ίσους κανόνες παιχνιδιού, ιδιαίτερα για πράξεις μεγάλου μεγέθους. Παρότι το κόστος μιας εκτέλεσης μιας πράξης μειώθηκε, το συνολικό κόστος για μια εντολή σε ορισμένες περιπτώσεις αυξήθηκε πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι κινεί τον επενδυτή και γιατί, ε, χρειάζονται, γιατί η MIFID παρακολουθεί ή όχι τις εξελίξεις στην αγορά. Επαναλαμβάνω, έχουμε όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές αγοράς και όχι μόνο για τις μετοχές, ακόμα και σε υβριδικά προϊόντα και σε παράγωγα και σε προϊόντα σταθερή απόδοση. Και εφαρμόζονται νέες εμπορικές στρατηγικέ πολύ μεγάλης ταχύτητας. 33.000 πράξεις το δευτερόλεπτο από ένα φορέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το 75% των πράξεων εκτελούνται από χρηματιστές και ενδιάμεσους. Πολλοί από αυτούς είναι σαν άτυποι δημιουργοί αγοράς. Δίνουν ρευστότητα χωρίς όμως τυπικές υποχρεώσεις. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις αγορές στο νέο αυτό οποίο. Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι να δώσουν τη δυνατότητα συλλογής κεφαλαίων και να βοηθήσουν τους επενδυτές. Παίζουν ένα βασικό κοινωνικό ρόλο οι αγορές είναι ισχυρές και αν υπάρχουν σημαντικοί εργαλεία που να μετατρέπουν το κεφάλαιο σε οικονομική ανάπτυξη. Όμως χρειάζονται οι ίδιοι κανόνες παιχνιδιού. Το ξεκίνησε αυτό η MIFID και εξασφαλίστηκε διαφάνεια και ισχύς στην αγορά. Η έκθεση θέτει ορισμένα σοβαρά ερωτήματα που εμείς ως νομοθέτη πρέπει να ανταλάβουμε υπόψη. Όπως όλα τα trading venues λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες. Δίνουν αξία και προστασία στους επενδυτές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι εποπτικές αρχές παρακολούν, είναι σε θέση να παρακολουθούν τους πάντες και, να, και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα venues Μπορούν οι ρυθμιστές μας να αποκαταστήσουν τα βιβλία ελέγχου audit books στην περίπτωση που συμβεί μια σοβαρή περίπτωση κατάχρησης στην αγορά. Συλλέγαμε λοιπόν όλα τα στοιχεία αυτά και ο κύριος λόγος στη δημοσίευση της έκθεσης που καθυστέρησε μέχρι τον Ιούλιο ήταν αυτός. Την περισμένη εβδομάδα είχαμε μια δήλωση ότι πολλοί θεσμικοί επενδυτές θεωρούνται ότι μεγάλα μεγέθη πράξεων θα οδηγήσουν σε αποχώρηση από την αγορά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από τα βροχυπρόθεσμα ωφέλη να μην υπονομεύσουν την στάση του συνόλου των επενδυτών. Και συμφωνώ με αυτό, γιατί η διάρθρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών μετά τη μύφη στην Ευρώπη προσφέρει πλεονεκτήματα. Μην γυρίσουμε το ρολόι πίσω σήμερα. Πρέπει όμως να υπάρξουν κανόνες και κριτήρια έτσι ώστε οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη να εξασφαλίζουν διαδίκες διαφανή βάση για τους επενδυτές, για όλους. Και με την έκθεση αυτή προσπαθούμε να λύσουμε ορισμένα από αυτά τα προβλήματα και ελπίζω η βοήθειά σας και η συμβολή σας να είναι σημαντική σε επόμενες Επειδή είναι πολύ τεχνική η έκθεση, Κάναμε και μια δεύτερη έκθεση, background, την κρατάω στο χέρι μου, σας τη δείχνω. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει και αυτή η δεύτερη που αναφέρεται σε τεχνικά θέματα, αλγορίθμους κλπ. Θα ακούσω τις απόψεις σας με πολύ προσοχή σήμερα και θα συνεχιστεί η δουλειά των σκιωδών παράλληλα με τη δική μου δουλειά έτσι ώστε ορισμένα βασικά διαθροτικά θέματα να αντιμετωπίσουμε σωστά και αυτό που πέτυχε η MIFID ω προ την ενιαία αγορά για όλους να είναι ένα ασφαλές δεδομένο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ Κέι. Ο Μάρκος δεν είναι εδώ. Έχουμε ποιους έχουμε από τους Τον κύριο Κάμπεν, Σιλβί Γκούλαρτ και Γιώργεν. Ο Γιώργεν είναι εδώ. Η Σιλβί πρώτη. Ε, εξ ονόματος Τόλε Σμιτ. Ευχαριστώ. Ο Σμιτ ε, ήταν σκιώδης. Ε, ε, μου ζήτησε, επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ λόγω της ε, εκστρατείας στη Σουηδία, μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Να πω καταρχάς ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε όλα τα σημεία. Βέβαια, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον Όλε. Επίσης θέλω να πω ότι το έργο της εισηγήτριας και οι βασικές κατευθύνσεις της μας βρίσκουν σύμφωνους αύξηση της προστασίας των επενδυτών, σημαντικό συγχρόνως οι των πιστοτικές υπηρεσίες να υποστηρίζουν την οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλό αυτό, φιλόδοξη, άρτια, ισορροπημένη στην προσέγγιση έκθεση, αλλά έχουμε ένα ερώτημα. Δεν νομίζουμε ότι πάντοτε απαντά ξεκάθαρα σε ερωτήματα που είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Παραδείγματο χάρη ζητάτε περισσότερη έρευνα ε, σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Και εμείς συμφωνούμε, πρέπει να διερευνηθούν ε, κάποια ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και τεχνικά. Αλλά ποιο είναι ακριβώς ε, το πεδίο, η εμβέλεια αυτών των ερευνών και ποιος θα είναι αρμόδιος για μια τέτοια διερεύνηση. Θέλετε τα κράτη-μέλη να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες στην Κομισιόν. Ποιος θα ήταν ε, ο ρόλος της ΕΣΜΑ και του ESRB, των δύο νέων δηλαδή φορέων. και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη τεκμηρίωση από τι τεχνικέ συμβουλέ που ισχύουν μέχρι τώρα. Σε ό,τι αφορά το συστημικό κίνδυνο, πράγματι ε, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα στο πλαίσιο τη αναθεώρηση τη οδηγία MIFID, αλλά θα πρέπει η MIFID να αναθεωρηθεί ώστε να παρέχει και περισσότερη προστασία στου καταναλωτέ και άλλου ε, στόχου που δεν έχει ακόμα εκπληρώσει. Υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα θέματα, μερικά στοιχεία μπορώ να σα δώσω τώρα. Θέλετε να μειωθεί το χρονοδιάγραμμα για τις διάφορες διαπραγματεύσεις και τη δημοσίευση, νέες διατάξεις ε, της ΜΥΦΙΤ παράγραφος 6 για τα δίκτυα διασταύρωση εντολών, τα BCN. Είναι δύσκολο αυτό. Ε, χρειάζεται να γίνει κάτι βέβαια, αλλά φοβόμαστε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της διαφάνειας. Και ένα άλλο τεχνικό σημείο πώς θα γίνει αυτή η μεταφορά από τα BCN, δίκτυα διασταύρωση εντολών, στα MTF, δηλαδή τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης. Κατά τα λοιπά σας ευχαριστούμε για την έκθεση. Θα δούμε τι θα ενταχθεί στην αναθεώρηση της MIFID και τι θα πάει σε άλλα πλαίσια. Αυτά είχα να πω προς το πάνω. Ευχαριστώ. Thank you, Sylvie. Um, I will ask the e Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι ασχολήθηκε με αυτό το δύσκολο θέμα και θεωρώ ότι μας παρουσίασε μία πολύ καλή επισκόπηση του συνόλου η οποία πρέπει να μας απασχολήσει ιδίω ε, εάν ε, πρέπει να εξετάσουμε πώς θα βελτιώσουμε και θα αναθεωρήσουμε ε, την Μίφιντ. Βέβαια ένας από τους λόγους του κακού είναι ε, και αναγνωρίζεται στην έκθεση ότι κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη και για να εξετάσουμε όντως το πρόβλημα σωστά πρέπει να το κοιτάξουμε από όλες τις κοπιές και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε μόνο ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τι θα μας προσφερθεί την Τετάρτη για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα διότι σε κάποιο σημείο, κάποια στιγμή πρέπει να λύσουμε αυτά τα θέματα. Ε, και εγώ σε ασυχία που έχω μέχρι στιγμής για τα παράγωγα δεν βλέπω καμιά λύση αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το συζητήσουμε και ίσως να περιμένουμε ως την Τετάρτη να δούμε τι θα μας δώσουν τότε. Ε, άρα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις συζητήσεις σε ε, άλλα θέματα. Επίσης ε, όσον αφορά τις λεπτομέρειες συμφωνώ με την συνάδελφο Γουλάρ Δηλαδή ε, ε, Μπορούμε, μπορούμε να δούμε ε, αν θα ενσωματωθούν οι νέες οργανώσεις ε, και πρέπει να δούμε κατά πόσον θέλουμε να να εμπλακούμε στα θέματα αυτά. Είναι θέματα που πρέπει να θυγούν. Ε, και θα πρέπει ίσως να ε, τα συμπεριλάβουμε στην έκθεση αυτή. Όσον αφορά τις ρυθμισμένες ε, αγορές, χρειαζόμαστε ενιαίους κανόνες για την ευρωπαϊκή αγορά ή μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει τώρα, δηλαδή η κάθε αγορά να καταρτίζει τους κανόνες της και ο συνάδελφος Σουίνβαν προτείνει να προβούμε σε ένα ε, stress test. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λύση, το συζητάμε, διότι ένα από τα βασικά σημεία είναι το ερώτημα εάν πρέπει να υπάρξουν ε, τιμές κατόφλια και μία διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων αγοράς. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα πεδία που τουλάχιστον από τη δικιά μου πολιτική ομάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια σκέψη εάν θέλουμε να διαφοροποιήσουμε τα μεμονωμένα θέματα ή να τα εξετάσουμε όλο συνολικά. Αλλά αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα στοιχεία που θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά τα όλα πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι ο συνάδελφος Σουίνμπερν έχει καταλάβει πολύ καλά την, ε, τη συλλογιστική αυτή και ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εικόνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κλούνερ ε, για τους σοσιαλιστές και όδης εισηγητής. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης εισηγητής ε, αντικαταστάτης ε, για τους σοσιαλιστές γιατί δεν μπόρεσε να παραστεί ο υπεύθυνος σήμερα. Θέλω να αναφερθώ εδώ στις ε, ε, σκοτεινές δεξαμενές και ε, την ενδιάμεση αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους κανόνες οι οποίοι αναφέρονται σε όλα τα θέματα μεταξύ των οποίων πρέπει να δούμε και την ανάγκη να αξιολογήσουμε τους κινδύνους διότι αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η διαφάνεια και η διαφάνεια θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις οικονομικές ανάγκες. Ε, βέβαια, το Κοινοβούλιο δέχτηκε τις ε, απαλλαγές και τις εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις, πράγμα το οποίο επιτρέπει να υπάρχουν αυτές οι σκοτεινές δεξαμενές και αποτελούν μία απειλή για τις χρηματαγορές. Η ρύθμιση των ε, αδιαφανών δεξαμενών τουλάχιστον θα λάβει υπόψη την ρευστή αξία και ε, θα μας επιτρέψει μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι το ποσοστό των συναλλαγών που γίνονται ανοιχτά ε, είναι 30 έως 40% και δεν καλύπτει τις επιταγές της ΜΥΦΗ γι' αυτό και ε, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν το ποσοστό το οποίο ε, το, το ποσοστό των συναλλαγών που διεκπεραιώνεται ανοιχτά έχει επηρεαστεί από τη μύφη και έχει μειωθεί. Ενώ ε, όσον αφορά τα δίκτυα και ε, τα, ε, τις συναλλαγές μέσω μεσητών βλέπουμε ότι αυτά είναι ρυθμισμένα όπως τα MTF και ε, ο εισηγητής τονίζει ότι πρέπει περισσότερες συναλλαγές να γίνονται εκτός των αδιαφανών δεξαμενών του OTC και να ε, εφαρμόζουν τους κανόνες της MIFID χωρίς να αποτελούν εξαιρέσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει δηλαδή να επιζητήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ε, να ε, ρυθμίσουμε τις απαλλαγές για να μην υπάρχουν ε, ζώνες αδιαφανείς στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Και τέλος πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι της ΜΥΦΙΝΤ εφαρμόζονται και στην πρακτική. Ευχαριστώ. Ο Πασκάλ. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι συμφωνώ με τα θετικά σχόλια των συναδέλφων για την έκθεση διότι πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο συζητήσεως υπησέρχεται και σε διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες και παρουσιάζει μια γενική θεώρηση η οποία μας ικανοποιεί και θα επιτρέψει να υπάρξει ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο που είναι απαραίτητη για να βαρύνει η φωνή μας στις συζητήσεις ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν η ΚΕΙ έλαβε το λόγο και είπε ότι η MIFID ήταν επιτυχία ήταν πολύ ευγενής διότι ο στόχος της MIFID ήταν να βελτιώσει τη διαφάνεια και περίπου όπως ελέγχθη 40% των, ε, ε, ε, των συναλλαγών γινόντουσαν over the counter δηλαδή ανοιχτά πριν τη MIFID και τώρα το ποσοστό παραμένει το ίδιο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγάλη ε, επιτυχία αυτή η ρύθμιση και πρέπει να υπάρξει μία βελτίωση ε, ουσιαστική και όχι απλώς επιφανειακή της ΜΥΦΙΤ. Ε, πιστεύω ότι συμφωνούμε με τις πρώτες προτάσεις της εκθέσεως διότι ε, αποβλέπουμε στην αύξηση της διαφανείας προ και μετά τη συναλλαγή και ίσως ε, κάτι το οποίο δεν καταλάβαμε καλά όσον αφορά την πρότασή σας για την βελτίωση της διαφάνειας είναι ότι θέλετε να κατεβάσετε το επίπεδο που θα επιμένει η συναλλαγές να διεξάγονται στα γνωστά dark pool. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε νέες συναλλαγές στο dark pool δεν θα βελτιώσουμε τη διαφάνεια, και ήδη αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα διότι οι ρυθμισμένες αγορές βλέπουν να απομακρύνονται ορισμένες και να αναχωρούν ορισμένες συναλλαγές στα μεγάλα κεφάλαια και η, τιμή που επιτεχάνεται εις τις ρυθμισμένες αγορές αντικατοπτρίζει όλο και λιγότερο το σύνολο των κερδών που γίνονται μέσω της συναλλαγής χ Οπότε οι αδιαφανείς δεξαμενές ε, των αγορών χρειάζονται μία τιμή αναφοράς και βασίζονται στην τιμή αναφοράς της ρυθμισμένης αγοράς. Εάν λοιπόν αυτή η τιμή δεν αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία των συναλλαγών ε, έχουμε πρόβλημα και αιτιολογήσεως της τιμής και επιτεύξεως των στόχων μας και των στόχων της MIFID που δεν επιτεύξησαν, δηλαδή δεν επιτρέπουν η τιμή η οποία εμφανίζεται στις ρυθμισμένες αγορές να είναι η δίκαια τιμή. Οπότε ε, η πρότασή σας ίσως βασίζεται σε μία έλλειψη κατανεωήσεως αυτής της ενίας. Το δεύτερο θέμα το οποίο έθιξε και ο κύριος Φέρμπερ ή η η σιλβη Γκουλάρ είναι να λάβουμε υπόψη τον ε, ρόλο της ΕΣΜΑ περισσότερο από ό,τι ε, προβλέπεται στην έκθεση διότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να καταρτήσει κοινούς κανόνες για όλες τις ευρωπαϊκές οντότητες. Υπάρχουν δύο ανταγωνισμοί, αφενός ο ανταγωνισμός στα πλαίσια των γνωστών και ίσων κανόνων για όλους και ας κερδίσει ο καλύτερος, χωρίς πρόβλημα. Και υπάρχει και ο ανταγωνισμός βάσει των κανόνων και αυτό είναι επικίνδυνο διότι δημιουργούνται ορισμένα προνόμια ή αντιστρόφως υπάρχει μία τάση για αρνητική, ε, ε, μία αρνητική πτωτική πορεία. Οπότε πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι οντότητες ε, τσακώνονται σχετικά με τους κανονισμούς και η ΕΣΜΑ θα είναι καλύτερη εποπτική αρχή από ό,τι εμείς αρχικά θέλαμε να υπολογίζουμε. Όσο τώρα για, το, για τις συναλλαγές δεν βλέπουμε πραγματικά γιατί οι μικρές επιχειρήσεις και η πραγματική οικονομία, το σύνολο των επενδυτών και όχι αυτοί αυτούς που κάνουν ήδη το high efficiency trading ποιο θα είναι το όφελος από αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει ακόμη να αξιολογήσουμε τις αιτίε για τις οποίες ε, γίνονται αυτά, αλλά η οδηγία δεν προσπαθεί να κατευθύνει τα πάντα, αλλά θα μπορούσε παραδείγματο χάρη να αφισβητήσει το γεγονός ότι το high frequency trading δημιουργεί μεγαλύτερη ρευστότητα. Ε, δηλαδή, ε, πιστεύω ότι ορισμένοι ρυθμιστές το λένε και ανοιχτά. Εάν ε, οι περισσότερες από τις εντολές οι οποίες ε, ε, γίνονται υπομορφήν high frequency trading είναι δοκιμαστικές και δεν υλοποιούνται τότε απλώς δοκιμάζουν την αγορά και δεν πρόκειται για ουσιαστικές συναλλαγές. Εάν λοιπόν απλώς εξετάζουν την αγορά και είναι προσβάσιες μόνο σε μια μικρή μερίδα και δημιουργούν ένα ολιγοπόλιο δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις μεθόδους. Ε, είμαι αρνητικό. Μία πρόταση θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε θα ήταν τουλάχιστον να ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες στα χρηματιστήρια να εισάγουν και να υποχρεώσουν τις εντολές οι οποίες καταγράφονται να χρεώνονται. Ενώ τώρα οι εντολές οι οποίες κατατίθενται και δεν εκτελούνται δεν χρεώνονται. Οπότε ε, θα μπορούσαν ε, όλα τα χρηματιστήρια της Ευρώπης να είναι υπό την εποπτεία της ΕΣΜΑ και να υπάρχει μία ελάχιστη τιμολόγηση για όλες τις εντολές οι οποίες κατατίθενται, πράγμα το οποίο θα ήταν πιο θετικό από την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ο σχιώδης εισηγητής της πολιτικής μας ομάδας είναι ο Τόμας Χέντελ, δεν είναι εδώ και γι' αυτό με παρεκάλεσε να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ε, ε, εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας και εκ μέρους του διότι ε, όταν κανείς ψάξει λιγάκι τι γίνεται και προσπαθήσει να δει τι συμβαίνει βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πηγές πληροφοριών. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο και γι' αυτό αυτό που έκανε η ΚΕΙ είναι πολύ καλό ότι προσπάθησε δηλαδή να θέσει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Επίσης, από μια διαφορετική οπτική γωνία εξετάσαμε να δούμε τι έχει γίνει στους τελευταίους μήνες όπου ασχοληθήκαμε με το Σοπροεβάζδορη package να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρηματαγορές και αν ε, εξετάσουμε τουλάχιστον από αυτό που κατάλαβα και διαβάζω σχετικά με τα dark pools ουσιαστικά συνέβη το αντίθετο διότι τα dark pools είναι οργανωμένη αδιαφάνεια. Οπότε το ερώτημα είναι, χρειαζόμαστε, υπάρχει κάποιο νόημα να επιτρέπουμε αυτά τα dark pools εάν αντιτίθενται σε αυτά τα οποία με τόσο κόπο προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τους τελευταίους μήνες ως προς το πακέτο εποπτείας. Δηλαδή πρόκειται για μία μορφή η οποία είναι τελείως αντίθετη σε αυτό το οποίο ε, προσπαθούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να απαγορεύσουμε τελείως αυτές τις μεθόδους διότι ε, επιτρέπονται από το 2007. Πριν το 2007 ζούσαμε μια χαρά χωρίς τα dark pools στην Ευρώπη. Άρα μήπως θα ήταν λογικό αυτές οι μορφές συναλλαγών να απαγορευτούν τελείως. Οπότε και εμείς ε, τότε ε, θα συμπεριφεθούμε κατά την ψηφοφορία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ε, υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή διότι δεν αποβλέπει στο στόχο μας. Αυτά ήθελα να σας πω ουσιαστικά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω μερικά σημεία που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Το ένα αναφέρεται στην έκθεση και υπάρχει ένα ένας και από τη μεριά του συγγητή, της συγγήτριας, την μη διακριτική πρόσβαση. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει πιο γρήγορη πληροφόρηση αν έχει κανείς τα χρήματα να την αγοράσει. Αυτός δεν είναι ο ορισμός για μένα για το μη άνηση μεταχείριση. Δεύτερο, είχαμε αυτή την επέκταση με τις νέες τεχνολογίες, νέες τεχνικές και τρόπους ε, εμπορικής δράσης. Αυτά δεν αφορούν μόνο τη MIFID, αλλά είναι και η οδηγία για την κατάχρηση θέσεων στην αγορά. Το μελετάει αυτό ήδη η Κομισιόν και το συζητήσαμε και στις διαβουλεύσεις, αν γίνουν τέτοιου είδους χειραγωγικές δραστηριότητες που είναι ουσιαστικά ψευτοεντολές, αυτό εμπίπτει στην οδηγία κατάχρησης αγοράς με τις ποινές που προβλέπονται. Δεν γίνεται με τροπολόγηση της MIFID. Βέβαια ε, υπάρχουν και πολλές άλλες επιπτώσεις για τα θέματα αυτά. Πόσο περισσότερη διαφάνεια, παραδείγματο χάρη, χρειάζεται. Γιατί η διαφάνεια ενδεχομένως μπορεί να κάνει και ζημιά στην αγορά με την επίπτωση που έχει στις τιμές. Και θα πρέπει αυτό να το μελετήσουμε προσεκτικά για να βοηθήσουμε την Κομισιόν ότι θα κάνει την αναθεώρηση της MIFID, η εισηγήτρια και πάλι. Ευχαριστώ. Έχουμε μια βάση για ευρεία συνένεση εδώ μέσα, νομίζω. Είναι πολύ σοβαρή αυτή εδώ η δουλειά. Και η προπαρασκευαστική για την αναθεώρηση της MIFID του χρόνου πρέπει να καταλάβουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της αγοράς Μαθαίνουμε, έχουμε μάθει πολλά και θα ξεκουρθήσουμε να μαθαίνουμε βέβαια όσον αφορά την υποδομή για τη δραστηριότητα σε αυτό το μέτωπο. Ευχαριστώ και πάλι τη γραμματεία και όλοι όσοι μας βοήθησαν, ιδιαίτερα τους ρυθμιστές στα κράτη-μέλη και τη ΣΥΖΑ επίσης και όλους αυτούς φορείς από την αγορά οι οποίοι φροντίζουν όσο γίνεται και αυτοί να καταλάβουμε όλες τις έννοιες. Από τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα, εικάζω ότι ίσως χρειαστεί μια ομάδα για να αναπτυχθεί η έννοια της ενιαίας αγοράς και η έννοια της εποπτείας, της απλής και ενιαίας εποπτείας. Κάποιος ρώτησε να τα κάνουν το κράτη-μέλη ή να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι Βρετανής συντηρητικός, πιστεύω ότι είναι ο ρόλος της ΕΣΜΑ και ζητήθηκε από τον Σίζαρ να κάνει πολλές τέτοιες μελέτες, νομίζω ότι η νέα αρχή στην ΕΣΜΑ αυτή θα πρέπει να επιφορτιστεί με αυτό το έργο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, όπου ζήτησε το Κοινοβούλιο. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί και το πλαίσιο αναθεώρησης με εργαλεία πέραν των μετοχών, γιατί στηρίζεται ουσιαστικά στις μετοχές, γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες για τις μετοχές. Υπάρχουν όμως και δομές που μοιάζουν με μετοχές που και αυτές παίζουν στο παιχνίδι και αυτές πρέπει να τις δούμε προσεκτικά διότι όταν έχουμε ρευστέ αγορές ηλεκτρονικής μορφής δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εφαρμόζεται και να ισχύει και η και για αυτά τα προϊόντα και σημαίνω αυτό που είπε ο Μάρκος Φέρμπερ για τα παραγωγά θα έχουμε το τελικό έγγραφο σε λίγο για να δούμε πού χρειάζεται να καλυφθεί περισσότερο η διάσταση παραγόγων και τα εργαλεία παραγόγων να υπόκεινται στο μέλλον στη MIFID για τα stress test. Με βάση τις τεχνικές πλατφόρμες που έχουμε, πολλά από χρηματιστήρια είναι πολύ εκλεπτισμένες τα έργα πλατφόρμες και μιλάμε για αξία 860 δις δολαρίων δηλαδή που εξαφανίστηκαν μέσα σε λεπτά στις Πολιτείες. Μπορεί να ανακτούν την αξία αυτή μετά από 25 λεπτά, αλλά πάρα πολλοί επενδυτές έχασαν πάρα πολλά λεφτά. Ενώ είχαν συγκεκριμένες στρατηγικές, προνοητικές, stop order κλπ. Και χάθηκαν τεράστια αξία από τα χαρτοφυλάκια των χρηματιστών λόγω ενός τεχνικού λάθους στη συγκεκριμένη μέρα. Πολύ προσοχή λοιπόν μην έχουμε τεχνικό βομβαρδισμό εντολών. Αυτό το λένε, το αποκολούν staffing. Υπάρχουν ένα σωρό ορολογία που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Αυτό το staffing σημαίνει ότι πέφτουν πάρα πολλέ εντολές και εκτελείται μόνο μία από μερικές εκατοντάδες. Χρειαζόμαστε συστάματα που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, να μην καταραίει η αγορά. Ίσως χρειάζονται και προδιαγραφές και πρότυπα έτσι ώστε να αντέχουν τα συστήματα όταν βομβαρδίζονται από τεράστιο αριθμό εντολών. Διαφάνεια. Συμφωνώ. Αν η αγορά λειτουργεί σωστά, θα κινούνται οι άνθρωποι με βάση πληροφορίες που έχουν προς τη πιο σωστή κατεύθυνση. Στις πιο φωτεινές αγορές, ας το πούμε. Να είναι πιο ελκυστικές οι αγορές και να μην χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το βούρδολο και το μαστίγιο ως κίνητρο. Πάντως θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό και στις επόμενες εβδομάδες περαιώνουμε το εξή. Δεν λέω ότι οι dark pools, οι διαφωνίες δεξαμενές είναι άχρηστες. Λέω ότι χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες, ιδιαίτερα για τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, να δρούνε με διαφάνεια πριν από την πράξη και να τις χρησιμοποιούν ο κόσμος όταν χρειάζεται και όχι σαν μια κλασική λύση ρουτίνας. Διαφάνεια λοιπόν, διορθωτική ε, ισορροπία στην αγορά, αναθεώρηση της MIFID και την αναθεώρηση της MAD, η οποία και αυτή θα γίνει στο, μέχρι το τέλος του χρόνου. Το είπα και στην αρχή. Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο και τον Μάιο με ένα θέμα πολύ επίδικο όσον αφορά τις ερωτήσεις που θέταμε σχετικά με την υψηλή συχνότητα πράξης, αδιαφωνίες δεξαμενές κλπ. Κρίνοντας από τα σχόλια και από την αγορά ε, της Ασίας και των Πολιτειών είμαστε μάλλον κλασικοί στη λύση μας. Και ελπίζω, όπως είπα, να εξασφαλίσουμε ευρεία συνένεση της επόμενης εβδομάδας. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε και 27 Σεπτεμβρίου όριο τροπολογιών. 8 Οκτωβρίου θα συζητηθούν. Στις 26 θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και θα περάσουν στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Πλησιάζουμε την ψηφοφορία. Παρόλα αυτά ας περάσουμε στο 5 διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων. Γνωμοδότηση Γιάνν Έπινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται οι αξιολογήσει των επιπτώσεων να είναι αντικειμενικέ. Στην γνωμοδότησή μα, λοιπόν, ουσιαστικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση επιπτώσεων από τον πρόεδρο τη Επιτροπή και ενό πάνελ από αξιωματούχου διαφόρων γενικών διευθύνσεων δεν εγγυάται την ανεξαρτησία ή τουλάχιστον πρώτης όψης δεν την εγγυάται. Επομένω η γνωμοδότησή μα έχει ως στόχο να τονίσει ότι είναι απαραίτητος εξωτερικό έλεγχος, κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. Ζητούμε λοιπόν να υπάρχει μία, ένας ανεξάρτητος ποιοτικός έλεγχος μετά από την παρουσίαση της γνωμοδότησής μου είχα κάποιες τροπολογίες, από τον κύριο Τόμας Μαν όλες, τις δέχομαι, τις δέχομαι στο σύνολό τους. Το μόνο που θα άλλαζα θα ήταν σε κάποια σημεία τη διατύπωση. Πάντως με όλες τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είμαι σύμφωνος και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος το λόγο. Έντουαρτ. Και πάλι εκπροσωπώ το σκιώδη συγκητή που δεν παρίσταται και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Γνωρίζουμε ότι επιτελέστηκε πρόοδος τα τελευταία πέντε χρόνια από την Επιτροπή για την Αξιολόγηση Επιπτώσεων. Αξιολόγηση Επιπτώσεων είναι ένα σημαντικό κομμάτι του όλου προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πιθανές επιπτώσεις πριν τη λήψη μια απόφαση, Βέβαια υπάρχει ακόμη δυνατότητα να ενισχύσουμε σημαντικά τη διαδικασία τη εξολόγησης των επιπτώσεων. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Σημειώνουμε επίση ε, την ανάγκη να υπάρχει δίκαια ισότιμη πρόσβαση για θελοντικέ ομάδε, για μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, που αγωνίζονται να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές, ανεξάρτητες ε, αξιολογήσεις επιπτώσεων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια εξωτερική τη όλη διαδικασία, γιατί αυτό θα ενίσχυε την ολιστική φύση, τον ολιστικό χαρακτήρα μια αξιολόγηση επιπτώσεων, ενώ εμεί θέλουμε να ληφθούν υπόψη και οι οικονομικοί παράγοντε, αλλά και οι περιβαλλοντικοί και οι κοινωνικοί παράγοντε. Με την ανάθεση σε εξωτερικό φορέα υπάρχει ο κίνδυνος αποσύνδεσης από τη διαδικασία αξιολόγηση επιπτώσεων και δεν θα υπάρξει επαρκής ε, προσέγγιση με τους ενδιαφερόμενους, τους ενδιαφερόμενους φορείς. Άρα θα αποδυναμωθεί η δυνατότητα του Κοινοβουλίου για αποτελεσματικό έλεγχο της νομοθεσίας. Τέλος, δεν συμφωνούμε ότι σωστή αξιολόγηση μπορεί να παρακολλήσει κάποιες φορές ε, τις ε, διαδικασίες και ότι θα πρέπει να γίνεται πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά το γάμα και τις παραγράφους 3 και 4 θα τις καταψηφίσουμε γιατί στόχος μας είναι να έχουμε άρτιες και αποτελεσματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Έπινγκ ο συντάξη γνωμοδότη θέλει να απαντήσει, να πει κάτι παραπάνω. Όχι, δεν σχόλιο κύριε Πρόεδρε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρο. Για να γυρίσω σελίδα λοιπόν και εγώ. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 28 Σεπτεμβρίου. Η Καθήλυνα Αρμόδια ψηφίσει τον Οκτώβριο, άρα η εκθέση θα συζητηθεί στη δεύτερη σύνοδο της Ολομέλειας του Νοεμβρίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 συζήτηση τροπολογιών επιστικής μου έκθεσης για την επιστροφή του φόρου προστέμενης αξίας. Αφού δεν υπάρχουν τροπολογίες δεν χρειάζεται να γίνει και συζήτηση. Το είχα πει και στις ανακοινώσεις του Προέδρου, της Προέδρου. Οπότε φτάνουμε στην ώρα των ψηφοφοριών. Πέντε λεπτά νωρίτερα τους είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε στις 6 παρα 25 λόγω του σημείου που προσθέθηκε στην ημερήσια διάταξη για την εποπτεία. Ερωτώ λοιπόν, μέχρι να μοιράσουμε τον κατάλογο των ψηφοφοριών, θα έχει έρθει ρώτο ή άλλος αλλά τι λέτε, ε, να διανύμω από τώρα τον κατάλογο των ψηφοφοριών, να δεν και η πρόεδρος ίσως και αυτή έναν κατάλογο. And have, have, have members... Έχετε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας, γιατί θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχω να σας εξομολογηθώ κάτι κυρία Πρόεδρε. Ξέχασα την κάρτα μου στο Στρασβούργο. Πρόεδρος, και εγώ το ίδιο, αλλά έτρεξε και την έπιασε και την πήρε ο βοηθός μου. Λοιπόν, κανένας άλλος που έχει ξεχάσει την κάρτα του. Μπορούμε να μετράμε και χέρια. Και αυτό γρήγορο είναι. Πάντως καλό είναι να μετράμε. Έχετε όλοι τους ε, καταλόγους ψηφοφορίας. Ας κάνουμε έναν έλεγχο. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε, είστε όλοι ικανοποιημένοι. Ωραία, 24 είναι χαρούμενοι, οι 8 δεν ξέρουν τι είναι. Πάντως το σύστημα δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Πριν περάσουμε όμως στην ψηφοφορία, θα έχουμε άλλα λίγα λεπτά, γιατί ο εισηγητή θέλει να μιλήσει πριν αρχίσει η ψηφοφορία και έρχεται τρέχοντα προς τα εδώ ο κύριο Μπούλμαν. Α, κύριε Κάρα. Κυρία Πρόεδρε, ε, ζητάω το λόγο για να σας βοηθήσω να κρατήσετε και να σεβαστείτε το, το χρόνο της ώρας των ψηφοφοριών και να βοηθήσω και τον κύριο Μπούλμαν που έρχεται. Έχω να πω τα εξής. Ωραία. Λοιπόν, Καταρχήν με ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι γιατί ψηφίζουμε σήμερα εφόσον η Επιτροπή της Βασιλείας συνεφώνησε εχθές. Ε, μπορώ να πω ότι χαίρομαι που σήμερα ψηφίζουμε διότι έτσι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεικνύουμε με ε, μία προσωρινή συμφωνία στη Βασιλεία 2 ε, ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας συνειδητοποίηση και από την άλλη πλευρά με την ψηφοφορία αυτή ε, να ε, ε, πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χωρίς προκαταρτική εργασία από τη δικιά μας Επιτροπή δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το προσωρινό αποτέλεσμα ε, της Επιτροπής Βασιλείας 2. Όσον αφορά τη Βασιλεία 3 και την συμφωνία πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μία προσωρινή συμφωνία μεταξύ εκπροσώπων τραπεζών διότι η ε, Βασιλεία 3 δεν είναι σε αυτό το στάδιο κάτι το οποίο είναι νομοθετικά δεσμευτικό. Όσον αφορά την αρμόδια επιτροπή για τη Βασιλεία δεν υπάρχει καμιά δέσμευση διότι 21-22 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί ακόμη το λεπτό θέμα του ορισμού της ρευστότητος και τρίτον μία απόφαση δεσμευτική για την Ευρώπη λαμβάνεται όταν οι Υπουργοί Οικονομικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει επί της οδηγίας. Είναι ένα βασικό στάδιο για μία σημαντική πρόταση την οποία επεξεργαζόμαστε αλλά στην έκθεση ακόμη υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Δηλαδή μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει συσσωρευτική μελέτη όλων ε, των ρυθμίσεων για τις τράπεζες οι οποίες είναι υποσυζήτηση δηλαδή ε, την απόσυρση των δημοσίων πόρων από την τράπεζα μόλις εφαρμοστεί η Βασιλεία 3. Επίσης η συζήτηση σχετικά με την κεφαλαϊκή επάρκεια ε, όπου συζητάται συγχρόνως η φορολογία των συναλλαγών και όλες οι συσσωρευτικές επιπτώσεις των ε, ευρωπαϊκών ρυθμίσεων θα πρέπει να διερευνηθούν κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μία σοβαρή αξιολόγηση των μέτρων και των ε, ε, εμπλοκών τους. Τρίτον, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ε, μελέτη της αποτιμήσεως των επιπτώσεων με τους αριθμούς οι οποίοι οδήγησαν εχθές σε μία προκαταρκτική συμβολία στην Επιτροπή για την Βασιλεία. Επίσης όσον αφορά τις τράπεζες και ε, τα κράτη που συμμετέχουν στην Επιτροπή της Βασιλείας συζητείται η αύξηση κατά 1% της κεφαλιακής επαρκίας. Δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να στηρίζει τους αριθμούς οι οποίοι συζητήθηκαν εχθές και που να αντικατοπτρίζει την πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ακόμη ασαφές το θέμα του ορισμού του κεφαλαίου. Και αυτή τη στιγμή, το γράφουμε άλλωστε και στην έκθεση, αναφέρεται εις, ε, ε, προτιμά την ε, προώθηση των πιστώσεων από την αγορά από την προώθηση των πιστώσεων από τράπεζες. Επίσης δεν υπάρχει καμία σύγκριση των Αμερικανικών ρυθμίσεων με τη Βασιλεία 2 και τη Βασιλεία 3. Εφόσον όλα αυτά δεν έχουν ε, ε, διευκρινιστεί και για να υπάρχει η ισότιμη ε, υποχρεωτική εφαρμογή των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών ρυθμίσεων θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει ότι δεν μιλάμε εδώ για εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής για τη Βασιλεία αλλά για ένα συντονισμό των οδηγιών διότι η σύγχρονη σύγχρονη εφαρμογή για την Βασιλεία με τις αμερικάνικες ρυθμίσεις είναι βασικό θέμα για τους Ευρωπαίους για να μπορέσουν να προωθήσουν τις επενδύσεις και την οικονομία στην Ευρώπη. Αλλά το, η έκθεσή μας συνεχίζει να είναι επίκαιρη και όσο υπάρχουν ακόμη πληγές και ανοιχτά θέματα πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Εμείς δεν μπλοκαριζόμαστε και θα πρέπει προσεκτικά και σοβαρά να ασχοληθούμε με αυτή τη συζήτηση. Προχωράμε το τρένο, αλλά υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν για λόγους σοβαρότητος και για λόγους διαφανείας. Ευχαριστώ τον τους σχεδιστές για την επικοδομητική συνεργασία της τελευταίας εβδομάδος, για τις συμβιβαστικές τροπολογίες και για την συζήτηση διότι η συζήτηση όσον αφορά ε, την ε, συμπεριφορά στις ε, μεμονωμένες τροπολογίες έχουν συζητηθεί λεπτομερώς μέχρι σήμερα το μεσημέρι αποδεικνύουν τις ανησυχίες θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και αν μέχρι τις 21-22 Σεπτεμβρίου συμβεί κάτι στο οποίο θα πρέπει να αντιδράσουμε έχουμε καιρό μέχρι μέχρι την Ολομέλεια 6-7 Οκτωβρίου να προβούμε σε τροπολογίες. Εάν παραμείνουν αναπάντητα ερωτήματα έχουμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τις κοινοποιήσουμε τις επιθυμίες μας όσον αφορά τα εκρεμή θέματα διότι είδατε ορισμένα πράγματα δεν αναφέρονται στην έκθεση διότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρομαι εδώ στις προτάσεις των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων. Θα πρέπει να ε, αναφερθούμε εις την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πρέπει να ενεργήσει. Και εφόσον όμως δεν έχουμε μέχρι στιγμής μία πρόταση και τώρα ξεκινά η εργασία μας δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Άρα ήταν σημαντικό να μην περιμένουμε το σχέδιο της ε, ε, οδηγίας αλλά να διατυπώσουμε μία έκθεση κατά τρόπον ώστε το Κοινοβούλιο πριν από όλους να αντικατοπτρίσει την κατάσταση της Βασιλείας στην ζωή μας και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην εφαρμογή της ρυθμίσεως αυτής. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ψηφίσουμε. Έχω στο κίτρινο εδώ γραμμένο τις οδηγίες της... Ε, Μου λέει γραμματεία, θα σα διαβάσω όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Your card 1. Παράγραφος το αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51, υπέρ, κατά, απογές. Παρακαλώ εδώ ηλεκτρονικό έλεγχο για την 51. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Αυτή ήταν η 51, η 52 κατά πίπτη, 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παρακαλώ να τα χέρια εμφανώς. Συμβαστική ε από πέντε ομάδες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική F σχεδόν όλοι είναι, συμφωνούν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική G από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5α64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική H τέσσερων ομάδων. Α, αυτή είναι, έχει τμήματα. Έχω μια, καταρχήν μια προφορική τροπολογία πρέπει να εμποδίζει τις ευρωπαϊκές αρχές να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη σταθερότητα του τραπεζικού κλάδου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος. Το πρώτο με την προφορική τροπολογία. καταπίπτει 19-19. Χωριστή ψηφοφορία ζήτησαν οι πράσινοι το πρώτο τμήμα. Είναι το σύλλογο του κειμένου με εξαίρεση αυτό που ξεκινάει τη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά το υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. λέει, ε, έχει στα αγγλικά, however, ωστόσο. Αυτό εγκρίθηκε. Τρυπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία για το 7α του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική για το 7β του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η συμβαστική J τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία των πρασίνων για την παράγραφο 8α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα πέντε ομάδων σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική έλα σχεδόν όλοι συμφωνούν η γκοειδή, η πράσινη κλπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική μη πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται με 23-16. Συμβαστική εν τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές συμβαστική όμικρον σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα size υπέρ against abstentions that's carried Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές. Μερικές ομάδες ψηφίζουν δύο φορές. Παρακαλώ. Όχι φιλελεύθεροι, όχι, όχι. Την 105 ψηφίζουμε. εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική π, χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 114, 115, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ Α, έχουμε μια προφορική εδώ τονίζεται ότι η ποσοτική το και και μακρονομικές αξιολογήσεις μπορεί να υποδεικνύουν ότι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 αποσύρθηκε, 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 119 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 120 καταπίπτει 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική R. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές 128 ηλεκτρονικός έλεγχος. απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 καταπίπτει. 131 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος 133. Εγκρίνεται. 134 υπέρ Θέλετε να ξαναψηφίσουμε την 133, 133 ηλεκτρονικά ξανά. «22 υπέρ 15 κατά». Θέλετε και το 132. Η 132 είναι σαφής. Δεν γυρίζει πίσω. Δημιουργεί κακά προηγούμενα αυτό. 134 υπέρ. Κατά αποχές ασαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 134. εγκρίθηκε. Συμβαστική S5 ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 143 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος του δευτέρου τμήματος. Εμένα μου φάνηκε σα, σαφές. Εγώ αποφασίζω. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, το δεύτερο τμήμα της 143. Απορρίπτεται. Συμβαστική τα 5 ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά πίπτη. 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, όχι. 160 υπέρ, χέρια παρακαλώ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα παρακαλούσα να κάνουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική U τριών ομάδων σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές με βοηθάει αν σηκώνουν τα χέρια όλοι υπέρ κατά αποχές ευχαριστώ πολύ εγκρίνει το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά τα περισσότερα χέρια είναι κατά. Καταπίπτει λοιπόν. Δεν σηκώσατε τα χέρια, δεν μετριέται η ψήφο σας. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα λέει η πρόεδρος της ε, συμβαστικής γιου. Εγκρίνεται, εγκρίθηκε. Απλώς ήταν στην τεμπέλιδες να σηκώσει τα χέρια. 165 με προφορική τροπολογία. Καταρχήν ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται προφορική για την 21 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Β πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180, 178, 179 καταπίπτουν Όχι, όχι, θα τις ψηφίσουμε. 100, θα τις ψηφίσουμε. 178 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 185 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος στην 185 εγκρίνεται. Συμβαστική X. Πέντε ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά 189. ογδόντα Περιμένουν τους κατά, χέρια κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδώ έχουμε μία ψήφο μπλοκ. Σε μπλοκ. Okay, we have a complicated business on liquidity here. The first thing to be voted. Έχω ένα πολύ πολύπλοκο θέμα εδώ για την ε, μόχλευση. Καταρχήν έχουμε την προφορική τροπολογία των πασίνων. Να προσταθεί το take loan after κλπ. Πώς είστε υπέρ με την προφορική αυτή τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. I think 15, 13, 12 is worth checking, you know. Θεωρώ ότι εγκρίθηκε. Αυτό είναι το σύνολο του μπλοκ με την τροπολόγηση της προφορικής τροπολογίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Yes, yeah. So we now go to 210. 210. Υπέρ. 210 είμαστε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος της 220 απορρίπτεται 221 υπέρ κατά αποχές Νομίζω και αυτή απορρίπτεται, αλλά σας παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε λοιπόν 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 228 υπέρ κατά η 227 εγκρίθηκε αλλά δεν σηκώνται πολλά χέρια ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 228 εγκρίθηκε 229 υπέρ κατά Αυτά είναι γελία πράγματα, σας παρακαλώ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία 229. Right. Okay. voted. Εγκρίθηκε αυτή. 230 υπέρ κατά αποχές Αν μετράω τα χέρια σωστά, νομίζω εγκρίθηκε, αλλά περίεργες ψηφοφορίες γίνονται εδώ πέρα. Συμβαστική ζήταση έγινε 237 άτομα σπανιπέρ. κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τελειώσαμε αυτό. Τώρα έχουμε το ποσοστό μόχλευσης, το δίκτυ μόχλευσης. Α, αυτό έγινε. Άρα πάμε στο 239. Αυτό ήταν μάλλον για την ε, συντελεστή μόχλευσης. Το 237 που είπα γίνονται περίεργες πληροφορίες, θέλετε να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Τι θέλετε. Ψηφίσαμε, ηλεκτρονικά ψηφίσαμε. Απορρίπτεται λοιπόν. You sure you're pressing the right buttons? Είστε σίγουροι ότι πατάτε το σωστό κουμπί. Κάποιος κάτι έκανε στραβά, δεν ξέρω ποιος. 239 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 240 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 240 Εγκρίθηκε 241 καταπίπτει, 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.43 υπέρ. Δύο υπέρ. Κύριε Λούλιν, τι πρόβλημα υπάρχει. Δυστυχώς δεν άκουσαν οι διερμηνείς. Ε, Τα έχω χάσει κι εγώ κύριε Πρόεδρε. Τη 242 την ψηφίσαμε. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί ε, είμαι σε σύγχυση κι εγώ. Λοιπόν, 243 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 244 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Έτσι νομίζω. Το ΕΛΚ ε, από μόνο του δεν μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, συμβιβαστική ZD. Προφορική τροπολογία στην τελευταία παράγραφο. Ποιοι είναι υπέρ με την προφορική τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν η κατατμήματα ψηφοφορία και έχουμε τώρα το υπόλοιπο κείμενο. Όχι, τέρμα. Α, ήταν αντί αυτού, οκ, το κατάλαβα αυτό. Ευτυχώς που το κατάλαβα δηλαδή. 245 υπέρ. 254, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, περίεργη, ε, περίεργο το αποτέλεσμα. 254 ηλεκτρονικά. Κύριε Κάρας, έχετε κι εσείς ένα πρόβλημα. Εγκρίνεται. Κοιτάξτε, αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας, τι να κάνω κι εγώ. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ Συγγνώμη, πάμε πίσω στην προφορική τροπολογία για την ετολική σκέψη ΑΑ. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 7, στο ΑΑ νέο υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Νομίζω, αλλά θα το ελέγξουμε καλύτερα, γιατί ήταν αμφίροπο. Εγκρίνεται. Τελικά. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 9 παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στο Β, ψηφιπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, να ελέγξουμε τη 14. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία προφορική στο ΒΕ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο Γ ψηφίζουμε το πρωτότυπο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στο δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στο δέλτα α κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο. Προφορική τροπολογία στο ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στο G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο του ΙΤΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΣΥ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στο J εγκρίνεται. Τροπολογία 42 έχει καταπέσει, 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 κατά, έχει καταπέσει 49 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική τώρα ψηφοφορία για την τελική επί της έκτησης αυτής της 38 υπέρ και 2 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Κάρας. Και περνάμε τώρα στη δική μου έκθεση. Μάλλον δεν θα έπρεπε να προεδρεύω εγώ. Μία όμως τροπολογία υπάρχει. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Είναι σαφές νομίζω. Για, την, ε, για το ΦΠΑ ψηφίζουμε. Λίγες ψηφοφορίες μείνανε, κουράγιο. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει, δύο δεν έχουν ψηφίσει. Ε, εντάξει. Και τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα συνολικά, πάλι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα κατάφερα να κάνουν κι άλλο ένα να ψηφίσει. Λοιπόν, περνάμε τώρα, εγκρίνεται η έκθεσή μου, περνάμε στο σημείο 9. Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, όχι. Γιατί έχει διαγραφεί. Α, κατά πιπ. Πού πάμε. Αρχικό κείμενο παραγράφου 2. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πού πηγαίνουμε τώρα. Τροπολογία 16 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19 Οψ, συγγνώμη, πάμε πίσω. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο παράγραφ 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα, υπέρ, Μισό λεπτό, συγγνώμη, πάω πολύ γρήγορα. Έχουμε καταρχάς μία προφορική τροπολογία. All households και households. Ποιοι είναι υπέρ. Α, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική γιατί κάποιος ε, ετάχθηκε κατά. Άρα πάμε στην αρχική και η συμβιβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Και τώρα πηγαίνουμε στην παράγραφο 7α νέα με μια προφορική τροπολογία και είναι σύμφωνοι με την τροπολογία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, 3 αποχές. Αυτά. Διάφορα υπάρχουν. Όχι. Ελεύθεροι να φύγετε. Ευχαριστώ.